θα δείτε τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές χτες το απόγευμα. Κάνετε πολύ φασαρία σήμερα, λέει η πρόεδρος. Voilà, c'est mieux. Vous trouvez, pardon, les décisions de la réunion des coordinateurs οι αποφάσεις λοιπόν των ε, συντονιστών έχουν διανεμηθεί εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι τις μισή. οι αποφάσεις αυτές θα θεωρηθούν δεκτές. Ο κύριος Μπαρ δεν έχει. Α, μόλις τώρα τις ε, διανέμουν. Λοιπόν, ό,τι παρατηρήσεις έχετε, παρακαλώ μέχρι τις μισή έχετε χρόνο μέχρι τότε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να σας πω... Α, η κυρία Γκραπίνη, διαδικαστικό. Θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν έχω τον, την κάρτα ψηφοφορίας, οπότε ε, θα ψηφίσω δια της χειρός. Θα σας λάβουμε υπόψη, κυρία Γκραπίνη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες θα ήθελα να πω ότι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, προκήρυξε ε, την, το βραβείο νεοπαγών επιχειρήσεων ε, στον τομέα της κινητικότητας. Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν για την απονομή του συγκεκριμένου βραβείου θα υπάρξουν δέκα επιχειρήσεις οι οποίες θα χρηστούν ε, leaders στον τομέα της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Ε, πρόεδρος ε, είναι ή μάλλον με Κίνας ο κύριος Μαρτζελά ε, που είναι υπέρμαχος ε, της κοινή χρήση ε, των ιδιωτικών αυτοκινήτων και από, διάφορες άλλες πιστοτικ... από διάφορα πιστοτικά ιδρύματα. Στις 7 Δεκεμβρίου έκλεισε ο κατάλογος των υποψηφίων 500 startups ζήτησαν να πάρουν μέρος. Η απονομή θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες μετά από τις 5.30 θα σας ενημερώσουμε ανάλογα και υπάρχει και ένα μικρό βίντεο το οποίο κρατάει δύο λεπτά για να καταλάβετε πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται θα σας το δείξουμε. Λοιπόν, ε, η Ευρώπη προσπαθεί να βοηθήσει για μια ακόμη φορά αυτού του είδους επιχειρήσεις και θα αναδείξουμε λοιπόν τις ε, υποδειγματικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, να σας οδηγήσω στην πιο πεζή, αν θέλετε, δραστηριότητά μας από εδώ και πέρα, τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Je ferme le vote. C'est bien, on est un nombre suffisant. Τέλος λοιπόν, έχουμε φυσικά τον απαιτούμενο αριθμό, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις διαμεθοδιακές υπηρεσίες παράδοσης πακέτων. Άντερσον, η εισηγήτρια, ψηφίζετε. Madame Grappini, je vous regarde. Σας είδα, κυρία Γκραπίνη. Je ferme le vote. Πέρα στις ψηφοφορίες. Allez, je ferme le vote. C'est adopté avec plus 37 voix pour. ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια στην κυρία Άντερς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχετε ένα λεπτό σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και όλες τις και όλους όσους εν πάση περιπτώσει πήραν μέρος στην προετοιμασία του εγγράφου αυτού, εσάς Πρόεδρε, προεδρεύσατε του τελευταίου τριμερούς διαλόγου με πολλή αποτελεσματικότητα. Ελπίζω στην συζήτηση στην Ολομέλεια να πάρετε όλοι μέλο για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας. Allez, Καλώς περνάμε τώρα στη δεύτερη ψήφο. Έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου. Καλώς ορίσατε κύριε Μαρινέσκου. Είστε καλά, πώς πάει, όλα καλά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Γκραπίνη υπερψηφίζει. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, 38 υπέρ. Η έκθεσή σας λοιπόν γίνεται δεκτή. Κύριε Μαρινέσκου, συγχαρητήρια. Ναι. Thank Καθυστερήσαμε. Σας ευχαριστώ. Ο συντονιστής μου με υποχρέωσε να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά για τη βοήθειά σας. Να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης. Οι Σκιώδης ήταν ιδιαίτερα χρήσιμοι και εσείς η ίδια και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι not you. and Sven, Να ευχαριστήσω και τον Σβέν από τη γραμματεία. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Έως ότου καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με περίεργες ιστορίες στο Συμβούλιο για από δικής μας πλευράς. Αυτή που ήταν κατά, η χώρα που ήταν ε, περισσότερο κατά, στο τέλος ε, ψήφισε την πρόταση, τελευταία βέβαια. Ευχαριστώ πάντως όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου, το μήνυμά σας θα το μεταφέρω. Η επόμενη έκθεση για την κατάρτιση των οδηγών φορτηγών. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, βρήκε την κάρτα της και η κυρία Γκραπίνη. Πέρα της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, η έκθεσή σας ε, έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κύριε Λούντγκεν, θέλετε το λόγο. Είπε ευχαριστώ ο κύριος Πράγματι, είστε αποτελεσματικός, λέει η πρόεδρος. Συνεχίζουμε με την απαλλαγή του 2016. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εξωτερικές Υπηρεσίες. Λοιπόν, Μόντε, Φέρμπερ, καλημέρα σε όλους. Νταλούντε και Μέσνερ. Θα ξεκινήσω με την κυρία Μόντε και μετά με τον κύριο Φέρμπερ. Μετά ο κύριος Νταλούντε και μετά η κυρία Μέσνερ. Στη συνέχεια θα, πάρει το λόγο, θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές και όσοι επιθυμούν από τα μέλη. Στο τέλος θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μας δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία. Ξεκινάω όμως με την κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Περιμένετε λίγο κυρία Ντεμόντε. Όσοι θέλουν να βγουν να το κάνουν παρακαλώ ήσυχα. Πόσα λεπτά έχω στη διάθεσή μου, Πρόεδρε. Τουλάχιστον τρία λεπτά. Μιλάμε για την απαλλαγή τη σχετική με, τις, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εξωτερικές υπηρεσίες δεν είναι απλά θα έλεγα λογιστική η προσπάθεια αυτή, είναι περισσότερο πολιτική αξιολόγηση. Υπάρχουν κάποια λάθη σχετικά με τα επιτρεπόμενα επίπεδα, όπως ακριβώς είχε σημειώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βρισκόμαστε κάτω από το όριο υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ε, ε, ενημέρωσης όπως βγήκε από τις λογιστικούς ελέγχους που θα πρέπει να καλυφθούν και υπάρχει επίσης ε, η σχέση, ο λόγος ανάμεσα στις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις που εκτελέστηκαν που είναι χαμηλότερο από το απαιτούμενο ποσοστό. Συνεπώς λοιπόν και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πληρέστερη διαδικασία πληρωμών. Αυτό αφορά και το Horizon 2020 και το CEF. Επιστρέφω τώρα στο CEF, το Connecting Europe Facility δηλαδή, υποστηρίχθηκαν 452 προγράμματα στον τομέα των μεταφορών για 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για να ολοκληρωθούν τα TEN-T, όπως επίσης ε, και η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Υπάρχει επίσης και το κομμάτι το σχετικό με τα FACE. Εμείς έχουμε ήδη πει ότι δεν είναι σωστό τα χρήματα να προέρχονται από τα κεφάλαια για τις μεταφορές, από τις πιστώσεις, συγγνώμη, για τις μεταφορές. Πάντως υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Υπήρξαν χρηματοδοτήσεις για 3,64 δις ευρώ για ένα σύνολο 29 προγραμμάτων, 25 για τις μεταφορές και 4 τα πολυτομεακά προγράμματα. Θα πρέπει να υπάρξει όμως περαιτέρω πρόοδος και σε σχέση με το Περιφερειακό Ταμείο και σε σχέση με τη Συνοχή. Και δεν μιλάω μόνο για τα δίκτυα μεταφορών, επίγεια δίκτυα, αλλά υπάρχουν και προγράμματα και ταμεία εγγυήσεων που ξεκίνησαν από το 2016 για την υπευθυνότητα, έλεγχο ε, και διαφάνεια και για τα θετικά βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για την μεταρρύθμιση του συστήματος του δημοσιονομικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και το αίτημα περαιτέρω απλοποίησης έτσι ώστε να υπάρχει η λεγόμενη μονοαπευθυντική θηρίδα. Ε, όχι μόνο στις μεταφορές, ε, αλλά μιλάμε συνήθως για τις μεταφορές και όχι για τον τουρισμό. Το 17 διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει μια γραμμή ειδική για τις τουριστικές δραστηριότητες και αυτό δεν επιτρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα χρήματα τα οποία τίθενται στη διάθεση ε, αυτού του σημαντικού τομέα της οικονομίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελμόντε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ευθύ αμέσω. Ποιο θα ήθελε το λόγο ή μάλλον να ακούσουμε καταρχά όλου του εισηγητέ. Ωραία, εντάξει, καλύτερα έτσι. Άρα θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Φέρμπερ που θα μα μιλήσει για το shift to rail και για τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Κύριο Φέρμπερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομο ε, για τι δύο εκθέσει απαλλαγή, ε, δηλαδή την ε, shift to rail και την ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι πρέπει να εκφράσω τις ευχαριστίες μου με τους εισηγητές ε, γιατί ουσιαστικά ισχύουν τα περισσότερα από όσα είχαν πει οι προηγούμενοι εισηγητές ε, για ε, τον έλεγχο των λογαριασμών. Έχουν πάντως οι δύο οργανισμοί για κάποια πράγματα ακόμη να κάνουν. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό σιδηροδρόμων, βρίσκεται σε μία φάση ανάπτυξης, υπάρχει σχετική νομοθεσία, φαίνεται ότι είναι καλά προετοιμασμένος οργανισμός σε ό,τι αφορά τη φάση της προπαρασκευαστικής. Υπάρχει αυτή η ανακατανομή και ε, μεταφορά αρμοδιοτήτων και θα δούμε κατά πόσον όλα θα λειτουργήσουν ε, καλά και στο μέλλον. Θα ήθελα να πω ότι για τον Οργανισμό Σιδηροδρομών ε, μπορεί να υπάρχουν κάποια καλά ε, πρότυπα, έχουμε διπλά πρότυπα, αλλά δεν ε, υπάρχει καλή σχέση κόστους ωφέλους. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσει σε ένα πρότυπο και όχι σε δύο. Και έχει το πρόβλημα των διπλών εδρών, αυτό ουσιαστικά, της διπλής έδρας. Αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα διπλά πρότυπα, τα δύο πρότυπα και σίγουρα υπάρχουν αυτές οι νέες ε, αρμοδιότητες στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού πακέτου που θα πρέπει να αναλάβει ο οργανισμός σιδηροδρόμων. Εκτός από αυτά, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, τα 27,5-28 εκατομμύρια ευρώ, τον προϋπολογισμό, ουσιαστικά τα πήγαν καλά. Έρχομαι στη δεύτερη κοινή επιχείρηση, μάλλον στη δεύτερη απαλλαγή που αφορά όχι έναν οργανισμό, αλλά μια κοινή επιχείρηση, το Shift to Rail. Υπάρχουν κάποιες ομάδες ενδιαφερομένων, τα λέω κάπως ε, αφηρημένα. Ε, είχαμε να δούμε και τον ε, προϋπολογισμό αυτού του, αυτής της, κοινής, της επιχείρησης που ήταν γύρω στα 50 εκατομμύρια. βλέπουμε ότι ε, κατά 98% οι διοικητικές δαπάνες ε, ε, εκτελέστηκαν και γενικώ τα ποσοστά εκτέλεσης ε, είναι πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά αυτή η κοινή επιχείρηση θέλει να εφαρμόσει προγράμματα, δεν έχει δηλαδή να δημιουργήσει μια σημαντική δομή και ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι ήταν ρεαλιστικό το πρόγραμμα εργασίας διότι 100% εκτελέστηκαν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Τώρα η κοινή αυτή επιχείρηση Shift to Rail σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό πλέον είναι αυτόνομη και μπορεί να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της. Ε, χρειάζεται να υπάρξει κάποια εσωτερική ενοποίηση, ε, εδραίωση ε, της θέσης είχαμε ασκήσει κάποιες επικρίσεις πέρυσι βλέπουμε να παραμένουν τα ίδια προβλήματα διότι με τα επιχειρησιακά προγράμματα θέλουμε να λειτουργούν, να υπάρξει και αυτή η εδραίωση της δομής ε, και αυτές, ε, αυτά τα κενά που είχαμε παρατηρήσει τώρα που πλέον είναι αυτόνομοι αυτή και κοινή επιχείρηση θα πρέπει να καλυφθούν. Πάντως παρά ε, τα προβλήματα αυτά, εμείς συστήνουμε να δοθεί απαλλαγή στους εκτελεστικούς διευθυντές. Φαντάζομαι θα έχει το λόγο της και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέρμπερ. Το λόγο τώρα έχει κύριος ε, Νταλούντε για τον ΕΑΣΑ. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ψήφισμα συμπεραίνει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, γνωμάτευσε ότι όλες οι δραστηριότητες ήταν νόμιμες ε, και τυπικά σωστές, ο προπολογισμό εκτελείται ε, σωστά. Ε, ένα αυξανόμενο τμήμα του προϋπολογισμού προέρχεται από τέλη και χρεώσεις, ε, αντί για επιδοτήσεις. Ε, οπότε δεν θα χρειαστεί να αυξηθούν οι επιδοτήσεις σε αυτή την υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέσνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Είχα να ανέλαβα λοιπόν το ευχάριστο καθήκον να ασχοληθώ με την απαλλαγή αυτού του οργανισμού, Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Όλα είναι νόμιμα και κανονικά, χαίρομαι που μπορώ να το πω αυτό σε ό,τι αφορά ε, τις ε, λεπτομέρειες. Τώρα φυσικά θα ψηφίσουμε υπέρ της απαλλαγής. Ε, κάποιες λεπτομέρειες πολύ καλά ε, λειτουργήσαν τα πράγματα. Ποσοστά εκτέλεσης ε, γύρω στο 98% ε, είχε να ασχοληθεί με την ρήπανση των θάλασσών. Υπήρξαν κάποια δαπάνες, κάποια κονδύλια τα οποία δεν εκτελέστηκαν. Τα κονδύλια λοιπόν μεταφέρθηκαν στο 2016. Το θέμα είναι ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει και μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και επίσης για την δήλωση των παραλήψεων ή των δυσλειτουργιών για να είναι ασφαλείς οι υπάλληλοι οι οποίοι δηλώνουν τέτοια κρούσματα, τέτοια περιστατικά. Ε, όλα αυτά όμως έχουν γίνει και πιστεύω με υποδειγματικό τρόπο. Επίσης έχει αναπτύξει ο οργανισμός ε, το εργαλείο παρακολούθηση σε σχέση με τις ε, συστάσεις. Υπήρξαν συστάσεις που είχαν διατυπωθεί μέχρι το 2016 και οι οποίες όλες έχουν υλοποιηθεί και αυτά είναι θετικά. Επίσης ε, ενισχύθηκε εντολή του οργανισμού πέρυσι έχει αναλάβει συνολικά καθήκοντα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Ακτοφυλακή, Προϊκού Οργανισμού μάλιστα Αφήκης και Ακτοφυλακή. Ε, υπάρχει ε, μια συνέργεια σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών και του Frontex, αλλά και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Ελέγχου της ΕΦΚΑ. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. επίση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ε, πλατφορμών ε, offshore. Επίσης ανέλαβε καθήκοντα νέα ο οργανισμός. Καλή συνεργασία, ε, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό. Επίσης ότι αφορά τη στήριξη του θεματολογίου για τη μετανάστευση. Υπάρχει καλή συνεργασία όπως είπαμε το Frontex, αλλά ε, ήδη έχει συμφωνηθεί ε, ένα τριετές πλαίσιο επίπεδου εξυπηρέτηση, μια συμφωνία επίπεδου υπηρέτηση, αυτό είναι το 2016 και επίσης για τη θαλάσσια επιχείρηση έχουν συναυθεί ε, συμβάσει για παροχή υπηρεσιών επιτήρησης. Υπάρχει επίσης η δέσμευση για τη μείωση του 5% των θέσεων εργασίας. Ε, ε, πράγματι λοιπόν παγώσαν και ορισμένε θέσεις, τέσσερι λόγω των περικοπών. Ε, παρέμεινε ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων, 2,46, αλλά για το 2017 προβλέπεται αύξηση κατά 14 θέσεις λόγω της συνεργασίας με την υπηρεσία ακτοφυλακή. Εγώ είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένη για το πώ πήγαν τα πράγματα, οπότε σα συστήνω να υπερψηφίσουμε και να χορηγήσουμε απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μέσνερ. Κυρία Ντεμόντε, έχετε ξανά το λόγο για το πρόγραμμα ΣΕΣΑΡ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, αναφέρομαι στην υπηρεσία ΣΕΖΑΡ, είναι ένα σημαντικό μέσο για την ολοκλήρωση των εννέων ουρανών όπως λέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εφαρμογή του ΣΕΖΑΡ 2020 και γι' αυτό είναι δύο, σε δύο τμήματα ο προϋπολογισμός. Το πρώτο αφορά το ΣΕΖΑΡ 1 το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ενώ το ΣΕΖΑΡ 2 χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το Horizon 2020. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, υπήρξαν κάποιες διοικητικές προκλήσεις λόγω ακριβώς της κατανομής σε δύο τμήματα του προϋπολογισμού. Υπήρξε ένα χαμηλό επίπεδο πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις και νομίζω ότι σε σχέση και καθυστερήσεις στα προγράμματα. Υπήρξαν και κάποια επιπλέον ε, δυσκολίες ε, για τη διατύπωση των πληροφορικών προγραμμάτων και ο προϋπολογισμός ε, επιβαρύνθηκε κατά 14,5 εκατομμύρια. Αλλά για το ΣΕΖΑΡ 1 μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα προγράμματα ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική διατύπωση των διαγωνισμών για να υπάρξει περισσότερη απλοποίηση όπως επίσης και συντονισμός των προγραμμάτων επιδότησης. Σχετικά τώρα με τα drones και εδώ το ΣΕΖΑΡ ασχολείται με τα θέματα αυτά έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία στα πλαίσια του ΣΕΖΑΡ 2020. Η πρόταση λοιπόν είναι θετική και γι' αυτό το Κοινοβούλιο προτείνω να χορηγήσει την απαλλαγή. Σας ευχαριστώ κυρία Ντεμόντε. Επί του συνόλου λοιπόν τώρα των απαλλαγών θα δώσω το λόγο. Ε, πείτε μας για ποιες απαλλαγές μόνο θέλετε να σχολιάσετε. Κύριε Μαρινέσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι θα καταθέσω κάποιε τροπολογίε. σε ό,τι αφορά την ε, εκτέλεση των κονδύλων του ΣΕΦ που πήγανε από το που πήγανε στο ΕΦΣΙ, αλλά ένα μικρό τμήμα. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα εκεί ε, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί από εκεί δεν μεταφέρθηκαν κονδύλια. Θέλω να ξέρω ποια είναι η προσταμένη αξία για την ε, δαπάνη των χρημάτων αυτών, σε ποια έργα, θέλω το προπολογισμό, το ποσό και το λόγο. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια σημαντική πληροφορία. Και για το πολιετές μετά το 2020. Έκανα την ερώτηση και στον Επιτροπό Έτιγκερ γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται με αυτή τη σύμβαση μεταξύ Κομισιόν και Eurocontrol. Σε ό,τι αφορά το Performance Review Body. Ποια είναι η προσθέμενη αξία και πώς λειτουργεί αυτή η σύμβαση. Είναι αποτελεσματική και το Eurocontrol είναι επίσης αποτελεσματικό και αποδοτικό. Είναι ένας φορές διαχείρισης δικτύων και πολλά είναι τα χρήματα που δίνουν οι επιχειρήσεις στο Eurocontrol. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η DG Move θα πρέπει να ζώσει ένα χάρτη με αυτά τα έργα. Τι χρηματοδότησαν. Έχουμε ένα πλήρη διάδρομο ή λείπουν συνδέσεις που καλύφθηκαν ή υπάρχουν μικρές περιοχές στην Ευρώπη αλλά δεν ε, υπάρχει αποτελεσματικότητα γιατί είναι σε αυτές τι περιοχές. Για τι μεταφορές θα ήθελα να ξέρω τι έργα προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για το Δούναβι. Έγινε κάτι. Χρηματοδότησαν τα κράτη-μέλη κάτι που έχει να κάνει με, τη, με το μέτρο μεταφορών στη στρατηγική του Δούναβι γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Για το Σέζαρ τώρα, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα κοινή αυτή επιχείρηση. Το θέμα είναι η διατουργικότητα να υπάρχει. Τα σύστηματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα. Στο Νότο τα έχει αναλάβει μια διαφορετική εταιρεία σε σχέση με την εταιρεία που έχει αναλάβει το Βορρά. Δεν υπάρχει λοιπόν, διαλειτουργικότητα. Δεν θέλαμε κάτι τέτοιο από το Σέζαρ. Θα καταθέσω και για το Σέζαρ λοιπόν τροπολογίες. Γιατί και πάλι πρόκειται για σημαντικά ποσά. Και θέλω να ξέρω κατά πόσον το αποτέλεσμα είναι χρήσιμο. Για το ενίο του Ευρωπαϊκού Εθέρου, όπω πει Ζαμπέλ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Φόρστερ. Θέλατε το λόγο. Ναι. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τη δουλειά τους. Νομίζω ότι εξέτασαν τις λεπτομέρειες που πραγματικά χρειάζεται να εξεταστούν. Ίσως υποβληθούν κάποιες τροπολογίες, αν και από την ομάδα μας κανείς δεν ζήτησε να γίνει τροποποίηση. Θα το δούμε. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Μία ερώτηση. Ο κ. Μανέσκου φεύγει βέβαια, αλλά ε, έθιξε το θέμα της διαλειτουργικότητας. Ήταν πολύ σημαντικό. Ε, μίλησε για το βορρά και το νότο, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο ακριβώς πρόγραμμα μιλάει. Είπατε ότι υπάρχει θέμα διαλειτουργικότητας μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Ότι έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα, ε, άλλο στο Βορρά, άλλο στο Νότο. Για ποιο πρόγραμμα, για ποια υπηρεσία μιλάτε. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Να το επιβεβαιώσω, να ρωτήσω κι εγώ τους συνεργάτες μου κλπ. Αυτό. Αν μπορούσε να μας διευκρινίσει ο κ. Μαρινέσκου. Κύριε Μαρινέσκο, ζήτησα μια συνάντηση με, το, με του Σέζαρ για να μάθω τις λεπτομέρειες. Αλλά ήδη κάποιες εταιρείε μου το επιβεβαίωσαν. Τα συστήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με βάση τις ιδέες που ανέπτυξε το Σέσαρ και, τα, και κατασκευάστηκαν ενώ και στην πράξη υλικά δεν μιλούν μεταξύ τους. Συνήθως οι βόρειες χώρες αγοράζουν από την Ίντρα και οι νότιες από, το, από την Ταλής. αυτά τα δύο συστήματα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Πρόκειται για διαχείριση της ε, κυκλοφορίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκο. Κύριο Στέλιτσκα, καλημέρα σας. Έχω τρεις παρατηρήσεις νομίζω για, τον, για την έκθεση κυρίας Ντεμόντε. και μία ενδεχομένω που μπορεί να γενικευθεί. Παράγραφος 9. Εκφράζει την απογοήτευση για την σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων. κάτι που έφερε και μεγαλύτερη περιπλοκότητα στον προπολογισμό και αυτό μπορεί να υποσκάψει τον βαθμό της διαφάνειας. Ζητώ Συγγνώμη, μιλάτε πολύ γρήγορα από ό,τι μου λένε. Ζητώ συγγνώμη. Αν μπορείτε λοιπόν να φρενάρετε λίγο, να επιβραδύνετε. Ωραία, θα το κάνω, Πρόεδρε. Θα επιβραδύνω τον, τον ρυθμό μου, της ομιλίας μου, όχι τον υπόλοιπο ρυθμό του σώματός μου. Ε, ε, η 9, λοιπόν, σας είπα για, ποιο, για τι πράγμα μιλάει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ανησυχία της, ε, Επιτρο... Ε, της του Υπολογισμού κατά βάση. Ε, πολύ σωστό να εξετάσουμε τον αριθμό των χρηματοδοτικών μέσων που έχουμε, αλλά αν η παράγραφος 9 μείνει όπως έχει, ίσως χρειαστεί να υποβάλουμε μια τροπολογία. Διότι ζητούμε τις συνέργειες, ζητούμε οι συνέργειες να είναι μια ε, ένα σημαντικό στίχημα για μας και δεν θα ήθελα να το εγκαταλείψουμε. Παράγραφος 11. Για την αξιολόγηση του ΕΦΣΥ. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Είναι καλή ιδέα. Αλλά θέλω να κάνω μια πιο γενική παρατήρηση. Θα ήθελα να εστιάσουμε τις απαλλαγές μας με τρόπο, ώστε να αξιολογούμε όχι το κατά πόσον ξοδέψαμε, δαπανίσαμε το 99% του προπολογισμού, το 58%, αλλά για το πώς το δαπανίσαμε αυτό. Πώς μετρούμε, για παράδειγμα, ε, την καινοτομία ενός προγράμματος καινοτομίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε κάθε φορά τι πρόοδος έχει σημειωθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Θα πρέπει να προσπαθούμε να μετράμε την απόδοση ενός προγράμματος, την πραγματική απόδοση και όχι μόνο τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν. Τελευταία παρατήρηση, παράγραφος 13. Συμφωνώ με την κυρία Ντεμόντε. Ο αριθμός των σφαλμάτων 4,1% είναι πραγματικά ψηλός. Ε, εντυπωσιακά υψηλός θα έλεγα. Η απλοποίηση των μέτρων λοιπόν είναι απαραίτητη και όχι μόνο εδώ σε αυτή την έκθεση, σε όλες, αλλά πραγματικά απλοποιούμε και μετράμε μετράμε την, την απόδοση, την αποτελεσματικότητα αυτών των, της της γραφειοκρατικής απλοποίησης. Θα πρέπει οι απλοποίησεις να υπολογίζονται, να μετρώνται και να ποσοτικοποιούνται. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταλούντε. Ζητήσατε το λόγο, έτσι δεν είναι. Έχετε άλλες ερωτήσεις, ερωτήσεις για, τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες απαλλαγές μήπως. <laughs> Μου έγινε κάποια ερώτηση, μου απευθύνθηκε ερώτηση, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ah, ο κ. Κράμερ είναι στη λίστα, συγγνώμη. Ούτε ο κ. Κράμερ. Ποιος είναι τέλος πάντων. Μα δεν θέλετε το λόγο. Ο κ. Φαν Μίλτεμπεργκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την απαλλαγή της ΕΑΣΑ δεν συμφωνούμε με, την, με τον κύριο Σιγητή, τον κύριο Νταλούντε που λέει στην παραφού 7 ότι θέλει να δει αν μειώθηκε η ευρωπαϊκή επιδότηση. Η προστιθέμενη αξία της ΕΑΣΑ είναι τεράστια και γι' αυτό λόγο χρειάζονται καινούργιε και περισσότεροι πόροι. Μετά ε, δεδομένου του Brexit ε, το πλεόνασμα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για, αυτό, για την ομάδα που ασχολείται με το Brexit. τα δύο τρίτα του προπολογισμού χρησιμοποιείται για διάφορα προγράμματα και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την επιτήρηση ε, της εφαρμογής των κανόνων. Ε, θα υποβάλω μια τροπολογία λοιπόν για αυτή την έκθεση. Σε ό,τι αφορά το Σέζαρ, εξαιρετική έκθεση κυρίας Δεμόντε. Μιλάει για τα drones και την αντίστοιχη μελέτη. Είναι σημαντικό να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή πολιτική και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ποσά για έρευνα και ανάπτυξη. Κατά τα άλλα είναι καλή έκθεση, αυτό μόνο θέλω να πούμε, μια τροπολογία εκεί. Merci Σας ευχαριστούμε, κύριε Φαν Μίλτεμπουργκ. Ροτ. Uh, Ευχαριστώ. Δύο-τρία σχόλια σε ό,τι αφορά την κοινή επιχείρηση Shift to Rail. και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συντηροδρόμων και το Shift to Rail ε, με την πάροδο των ετών βελτιώθηκαν ε, σημαντικά, αυτό πρέπει να το πούμε, νομίζω. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό στηροδρόμων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι υπάρχει υψηλά ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων. 99% και 92% αντίστοιχα σε ό,τι αφορά ε, τον αίτησιο προβλησμό του 2016. Όμως υπάρχουν και κάποια σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου για το 95% το στόχο δηλαδή εκτέλεσης ε, των πληρωμών εντός ε, προθεσμίας 30 ημερών. Αυτό δεν κατάφερε να το κάνει ε, ο ΕΡΑ επειδή το ποσοστό των τιμολογίων που επεξεργάζονται τα μέλη, οι υπάλληλοι μέσα σε αυτό το ποσοστό των 30 ημερών δεν είναι υψηλό. Σημειώνω την παρατήρηση του κ. Φέρμπερ και αυτό που είπε και ο κύριος Φέρμπερ για τη διπλή έδρα από το 2013 είχε ζητηθεί να αλλάξει αυτό το διπλό καθεστώς, στα διπλά πρότυπα, όμως ε, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Ε, τα ξέρουμε και από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι γίνεται με τις έδρες, τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά το shift to rail, στόχος είναι να έχουμε μια, ένα νέο χώρο σιδηροδρόμου και εδώ έχουμε 100% ποσοστά εκτέλεσης για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Σημειώνω όμω και κάτι άλλο. Για τον επιχειρησιακό προπολογισμό, για τι πληρωμέ, ε, τα ποσοστά εκτέλεση ήταν λίγο χαμηλότερα. 86,6% και συνολικά 82%. Άρα εδώ θέλει βελτίωση. Η δε στρατηγική της Κομισιόν δεν έχει ακόμη θεσπιστεί. Και το ΣΥΦΤΟΡΙΛ πρέπει να βελτιώσει τη στρατηγική διαχείριση κινδύνου. Υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες του ελεγκτικού συνεταιρίου σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Αποφασίστηκε ε, πάντως να εφαρμοστεί μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό. Έχουν αναγνωριστεί αυτά τα σχόλια. Αυτά έχω να πω. Θέλω να ευχαριστώ τον Μάρκο Φέρμπερ για του δύο αυτού φακέλου πανέλα. Ευχαριστώ πολύ. Και αφού ακούσαμε τις ερωτήσεις, θα στραφώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Παρά, καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Τα σημειώσαμε πάντως. Και στα πιο ειδικά ερωτήματα θα απαντήσουμε γραπτός. Γενικά, με ικανοποίηση διαβάσαμε τα σχέδια έκθεσης που παρουσιάζουν τις επιτυχίες των οργανισμών αλλά και κάποια σημεία που χρήζουν βελτίωσης και χαιρόμαστε που η πρότασή σας είναι να χορηγηθεί απαλλαγή. Προς ενημέρωσή σας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια ομάδα εργασίας για την υλοποίηση μιας στρατηγικής εποπτείας ε, των οργανισμών, όλων των οργανισμών και ιδιαίτερα των ρυθμιστικών, για τις όποιες συστάμε σήμερα. Έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη και περισσότερο υπόψη και να υλοποιήσουμε συστήματα ελέγχου για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις αυτών των οργανισμών. Και επίσης να δώσουμε συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής σας. Επομένως, ε, νομίζω πως ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τις ε, εκθέσεις και όλα δείχνουν ότι το έργο των ε, οργανισμών αυτών που είναι και πολύ σημαντικό το, ε, την χάνει εκτίμηση γενικώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραμουμπάρ. Κυρία Ντελμόντε θα πάρει τώρα το λόγο. Θα συμφωνήσω να κάνω μόνο ένα σχόλιο για όλες τις εκθέσεις. Δέχομαι με ικανοποίηση τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, όπως είπα και εγώ στην αρχή, πρόκειται για πολιτικές παρατηρήσεις και όχι για καθαρά λογιστικές σχετικά με τις προτάσεις του συναδέλφου Μαρινέσκου. Συμφωνώ ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και περαιτέρω έλεγχη από πλευράς του Eurocontrol και σε σχέση με τα TNT, γιατί πάρα πολύ συχνά ε, υπάρχει ανάγκη να δούμε πού βρίσκονται τα προγράμματα και τα στάδια εκτέλεσής τους έτσι ώστε να υπάρχει ο σωστός έλεγχος σχετικά με τα ΣΕΣΑΡ και εγώ ε, είμαι υπέρ της διαλειτουργικότητας και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο τμήματα του συστήματος. Σχετικά τώρα με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Τέλιτσκα, αν υπάρχουν κάποιες ειδικέ παρατηρήσεις σχετικά με το καινοτομικό τμήμα, νομίζω ότι ο χώρος εδώ είναι κατάλληλος έτσι ώστε να αξιολογήσουμε αν η λογιστική διαχείριση της υπηρεσίας αυτής είναι η αναμενόμενη. Και τέλος, σχετικά με την διαδικασία απλοποίησης, θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε μια απλή ανακοίνωση και δημοσιοποίηση, αλλά να βρούμε ένα το κατάλληλο σύστημα για να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε και τίθεται γενικότερα το θέμα του στόχου των ευρωπαϊκών πιστώσεων. Δυστυχώς όταν δεν υπάρχει απλοποίηση ε, τα αποτελέσματα αργούν. Και για τον κύριο Βαν Μίλτεμποργκ για τα drones συμφωνώ ότι απαιτείται ε, περισσότερη διευκρίνηση του σημείου αυτού. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα κάποια κριτική για τον Οργανισμό Ασφάλισης Θάλασσα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να προκύψουν τροπολογίες ε, ε, και θα τις μελετήσω εφόσον ε, μου κατατεθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Φέρμπερ, ναι, ευχαριστώ πολύ. Η μία πολιτική ομάδα μιλά για ποσοστά εκτέλεση και ασκεί κριτικές και άλλοι... Ε, συνάδελφοι ε, λένε ότι ε, πρέπει να τα δούμε τα ποσοστά αυτά εκτέλεσης πιο συγκεκριμένα. Θα περιμένω τις σχετικές τροπολογίες. Εδώ για το shift to rail πρέπει να πω ότι δεν εξασφαλίζεται χρηματοδότηση μόνο από την Κομισιόν αλλά και από τι επιχειρήσει. Θα πρέπει και είναι σημαντικό να δούμε τι θέλει η βιομηχανία και τι είναι διατεθειμένη να πληρώσει γι' αυτό. Ε, ή μείναμε σε δηλώσεις προθέσεων και δεν είχαμε τίποτε στην πράξη. Αυτά τα αναφέρω και στη δική μου την έκθεση σε ό,τι αφορά ε, τις Συμφωνώ και εγώ και επαναλαμβάνω αυτό που είπε η συνάδελφος Μάισνερ. Περιμένουμε τις τροπολογίες για να τις μελετήσουμε για να έχουμε μια καλή έκθεση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Monsieur Έγινε ένα σχόλιο για την ενδεχόμενη μείωση της επιδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Εγώ απλώς είπα ότι ε, η υπηρεσία αυτή έχει ε, πλεόνασμα, οπότε εν ώψη του Brexit και εν ώψη του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει την ε, καλή χρήση των πόρων ε, της ε, θα μπορούσε αυτή η υπηρεσία να είναι υποψήφια. Δεν είπα ότι κάτι τέτοιο έχει αποφασιστεί. Κυρία Φώστερ. Μια διευκρίνηση, Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος, η Eurocontrol δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό σώμα, δεν αποτελείται μόνο από τα κράτη-μέλη και δεν χρηματοδοτείται αποκλειστικά από αυτά, αλλά από τα τέλη κυκλοφορίας των αεροσκαφών. Και το Eurocontrol δεν είναι η ΕΦΣΑ, είναι εντελώς διαφορετικό σώμα. Τα μέλη της Eurocontrol δεν είναι μόνο 28 χώρες. Το Eurocontrol είναι υπεύθυνο για όλες τις χώρες ΙΚΑΟ, 34 στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη διευκρίνηση. Το ΣΕΣΑΡ είναι άλλο πράγμα, η ΆΣΑ είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 25 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Καλώς, θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας με την έκθεση του κυρίου Ισμαήλ Έρτογκ για τις ε, παράνομες επεμβάσεις στα ταχύμετρα των ε, ε, επαγγελματικών οχημάτων. Προτάσεις για το αναθεώρηση του νομικού πλαισίου. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Έρτογκ, και μετά θα δώσω το λόγο στους Κιώδης και στα μέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα. Μιλάμε για την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιόμετρων. Ουσιαστικά αυτό αλλάζει παράνομα, μη εξουσιοδοτημένα, ε, τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ε, είναι ένα πολύ δεδομένο φαινόμενο στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο. Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ φθηνό. Δεύτερον, γιατί είναι κάτι πολύ απλό. Και τρίτον, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, θεωρείται ένα αδίκημα ε, όχι τόσο σοβαρό, δηλαδή δεν θεωρείται απάτη. Και έχουμε ε, αυτό το φαινόμενο στο 12% μεταχειρισμένων οχημάτων ε, στις ε, αγορές των κρατών μελών και διασυνοριακά μπορεί το φαινόμενο αυτό να εξαπλώνεται και να καλύπτει το 30 έως 50% των μεταχειρισμένων αυτή η παραποίηση δηλαδή των διανθέντων χιλιόμετρων και αυτό σίγουρα οδηγεί σε ζημία. Το είχαμε συζητήσει την τελευταία εβδομάδα της Επιτροπής που λάβαμε τη σχετική μελέτη 6 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ ε, είναι η ζημιά ετησίως από την παραποίηση των δεδομένων αυτών των ε, μετρητών. Και επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, ε, πλήττεται και η οδική ασφάλεια, πλήττεται και το περιβάλλον. Δηλαδή, εάν έχουμε παραποιήσει τα διανυθέντα χιλιόμετρα μπορεί να πάμε με καθυστέρηση στο συνεργείο για τον τεχνικό έλεγχο με αποτέλεσμα τα οχήματα να γίνονται λιγότερο ασφαλή συνολικά και όταν ε, τα διανυθέντα χιλιόμετρα έχουν παραποιηθεί αυτό ε, έχει να κάνει και με τις εκπομπές υψηλότερων ε, εκπομπών καυσαερίων και αυτό βλάπτει το περιβάλλον. νομίζω ότι το Βέλγιο ε, και η Ολλανδία έχουν αντιμετωπίσει με υποδειγματικό τρόπο το πρόβλημα. Υπάρχει το Car Pass System στο Βέλγιο και η Ολλανδία έχει ένα εθνικό σύστημα το Pass για την αποτροπή αυτών των παραποιήσεων. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό αυτό που κάνουν. Σημειώνεται δηλαδή ε, σε κάθε επίσκεψη συνεργείο ε, ο αριθμός των ενθέντων χιλιόμετρων ε, και, σε χιλιόμετρων και σε οποιαδήποτε άλλο τεχνικό έλεγχο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίηση. Στην Ολλανδία δίνει ο κατασκευαστή, ο αγοραστή μάλλον, το πιστοποιητικό ότι είναι σωστά τα χιλιόμετρα που αναφέρονται στο μετρητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει μιμητέ, ε, γιατί έχουμε συνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, ε, που είναι κάτι πάρα πολύ αναγκαίο θέλουμε να καταπολεμήσουμε το διοσυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων την παραπίση δεδομένων των μετρητών. Και εκεί πρέπει να ενισχύσουμε ε, τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως το CarPass και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους ειδικούς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που λέγεται ο Ρικάρις, Ιουκάρις, ε, η πλατφόρμα αυτή ε, και το πώς θα το κάνουν εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να αποφασιστεί ότι θα πρέπει να γίνει και σε κάθε έλεγχο, σε κάθε επίσκεψη στο συνεργείο μπορεί να μπει αυτή η εγγραφή στο, στην πλατφόρμα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό το μοντέλο γιατί είναι φθηνό, μπορεί πάρα πολύ σύντομα να εφαρμοστεί και είναι και απλό και βοηθά πάρα πολύ τους ε, καταναλωτές. Μπορεί να φέρει 8 δις ε, ετησίως. Δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με τεχνικές βελτιώσεις ε, ε, πράγματι δεν πηγαίνουν τακτικά στο συνεργείο όλοι οι οδηγοί τα αυτοκίνητά τους και σε ό,τι δεν αφορά τους βασικούς ελέγχους ε, ε, πολλές φορές δεν γίνεται αυτός ο έλεγχος εγκαίρος και υπάρχει αυτή η δυνατότητα παραποίησης του μετρήτη. Ο κατασκευαστής ε, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ε, ασφαλείς ε, τεχνικές. Υπάρχουν ήδη σήμερα αυτές οι τεχνικές, απλά θα πρέπει να τις εισαγάγουν γενικώ στα οχήματα. Υπάρχουν αυτά τα modules ασφάλειας, οι ενότητες ασφάλειας λογισμικού που δεν κοστίζουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Και με αυτές τις τεχνικές λύσεις μπορεί κανείς ε, βέβαια ε, είναι πιο ασφαλής, δεν μπορούμε να είμαστε 100% γιατί αυτό δεν υπάρχει. Αλλά σίγουρα μπορεί να βελτιώσει πολύ τα πράγματα. Και ε, θα γίνει πολύ πιο δαπανηρό για τους απατεώνες να παραποιούν τα δεδομένα των μετρητών. Άρα έχουμε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέσο το οποίο προτείνω και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει επιγόντως ε, να ε, προχωρήσουν στην των νομοθετικών μέτρων που θα χαρακτηρίζει απάτη την παραποίηση αυτών των δεδομένων των μετρητών. 26 κράτη-μέλη. Το 28 η παραποίηση είναι απαγορευμένη, αλλά μόνο σε 10 κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα για τους καταναλωτές ε, να μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα των μετρητών. Με τη βοήθεια λοιπόν των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ζητηθεί να υπάρξει συγκρίσιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη που θα έχει αναλογικές ε, κυρώσεις, αποτρεπτικές κυρώσεις για την παραποίηση αυτών των ε, φαινομένων. Και υπάρχει και το θέμα της συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας blockchain των αλυσίδων συστοιχειών. Και εδώ στρεφόμαστε στο μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας που δεν είναι και τόσο μακρινό. Είναι όλο και περισσότερα οχήματα συνδεδεμένα και ανταλλάσσουν δεδομένα. Ήδη λοιπόν σήμερα ε, υπάρχουν στοιχεία για την ε, μέση ταχύτητα, παραδείγματο χάρη, για την, ε, αλλά και για τα διανθέντα χιλιόμετρα. Με αυτή την τεχνολογία blockchain, που ουσιαστικά είναι μια τεχνολογία κρυπτογράφησης, είναι ασφαλής, είναι κεντρική και νομίζω ότι με αυτήν την τεχνολογία μπορεί να προσφερθεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους, και προστασία για τους καταναλωτές. Σήμερα ήδη υπάρχει ένα project, το Car Trust Chain, που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ασφαλή μέτρα, εύκολα μέτρα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Ήδη το κάνουν αυτό δύο κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ε, ανταλλαγή ε, δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε κάποιες ευρωπαϊκές ενιαίες ε, προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πολύ συναρπαστικά αυτό που μας είπατε κύριε Ερτούκ, πραγματικά συναρπαστικά κύριε Ερτούκ. Είπατε ότι υπάρχουν δύο κράτη-μέλη που ε, λειτουργούν υποδειγματικά. Μιλήσατε για την Ολλανδία και για το Βέλγιο. Αν κατάλαβα καλά και πραγματικά μας προκαλούν ήλικο τα στοιχεία που αναφέρατε. Είπατε 6 με 8 ε, δις απάτης ετησίως. 12% στο στόλο, ε, του στόλου. Και μιλάτε για τα με κινητήρα μόνο. Για τα φορτηγά έχετε στοιχεία. Εκεί έχουν τον ταχογράφο βέβαια, αλλά δεν ξέρω. Μήπως υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω η μελέτη σας αν έχει δώσει αποτέλεσματα και πάνω σε αυτά. Ε, τα φορτηγά λοιπόν και τους ταχογράφους. Είναι πολύ συναρπαστική αυτή η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μπαχ δυστυχώς έπρεπε να πάει να ψηφίσει σε μια άλλη επιτροπή, στο την κατανοησή σας. Έχω όμως ε, τη δήλωσή του και μπορώ συνοπτικά να πω και τα, τις δικές του απόψεις ε, και τις δικές μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο ε, Ερτούκ για την έκθεσή του. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και χρόνια ε, βλέπει κανείς και σε μεγάλους, ε, μεγάλα σωματεία αυτοκινητιστών ε, ή οδηγών να αναφέρουν αυτό το πρόβλημα. Ήδη από το 1990 υπάρχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες ψηφιακοί μετρητές. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να κάνει και κανείς τίποτα. Απλά γυρίζει πίσω το κοντέρ. Το λέω τόσο απλά και παραποιεί τα δεδομένα των μετρητών διενθέντων χιλιόμετρων. Ε, η κατασκευαστέ πρέπει να λάβουν τι ευθύνε τους και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέει και ο κύριο Ερτούγκα. Θα πρέπει και αυτοί να σκεφτούν τι γίνεται, ε, αν αυτό είναι δική του αρμοδιότητα, σε ό,τι αφορά δηλαδή και την ε, ε, ταξινόμηση των οχημάτων. Εγώ έχω μελετήσει αυτό το βελγικό μοντέλο εδώ και χρόνια, πραγματικά λειτουργεί καταπληκτικά, γιατί ανά πάσα χρονική στιγμή που γίνεται κάτι με το αυτοκίνητο, καταγράφεται και ο μετρητής. Τα δεδομένα του μετρητή δεν θέτουν χιλιόμετρων, είτε πρόκειται για επίσκεψη στο συνεργείο, είτε πρόκειται για τύχη το πρόκειται για έλεγχο ε, από την τροχέα. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ε, και είναι σχετικά καλή η ε, λειτουργία και περιορίζεται έτσι το ενδεχόμενο παραποίησης. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Έχουμε καλύτερο hardware, έχουμε καλύτερο σταχογράφους, όμως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα γιατί υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί hacker και πάρα πολύ ε, εύκολο είναι να υπάρξει ε, παραβίαση. Δεν είναι ένα απλό αδίκημα, ένα παράπτωμα. Η παραποίηση είναι απάτη και αυτό πρέπει να το πούμε. Ε, και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την τιμή τιμή ε, ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι τα χιλιόμετρα και όσο πιο λίγα τόσο πιο ε, καλά μπορεί να πουληθεί ένα αυτοκίνητο ε, και γι' αυτό δίνονται κίνητρα για αυτή την παραποίηση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν πενικό αδίκημα πάντως στην παραποίηση του δεδομένου των μετρήσεων. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με την πρόταση του Ισμαήλ. Και τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπαχ, ναι, πρέπει να τα σκεφτώ στα αγγλικά, τέλο πάντων ε, είναι πρόκληση αυτή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα περιοριστώ στο ότι η έκθεση ε, βρίσκει μεγάλη υποστήριξη από εμάς είναι μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους αγοραστές μεταχειρισμένων, τους καταναλωτές και χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, επιτέλους ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και θέλω να ασκήσουμε όλοι μαζί πιέσεις και στους κατασκευαστές που αναλάβουν τις ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Ο επόμενος ομιλητής έχει το λόγο. Ο κ. Σμάκερ. Ε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αρτού για τη δουλειά που έκανε. Όταν διάβασα το προσχέδιο είδα πολλά θετικά στοιχεία το ότι εστιάζει στα τεχνολογικά μέσα τις βάσεις δεδομένων και τα συνδυάζει προκειμένου να καταπολεμήσουμε την απάτη είναι πολύ καλά. Αλλά θα χρειαστούμε χρόνο, θα καθυστερήσουμε έτσι. Και θέλω να υπογραμμίσω τον επίγοντα χαρακτήρα αυτού του θέματος. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ σε απάτη η απάτη αυτή μας κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ταυτόχρονα τίθενται και θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος κλπ. Θα πρέπει να βάλουμε τέρμα σε αυτό το φαινόμενο. Το συντομότερο. Θα πρέπει το σύστημα που θα εφαρμόσουμε να είναι εύκολο και να, να μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να έχουμε βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ. Ήδη έχουμε το ή Ιουκάρις. Το Βέλιο, για παράδειγμα, συνεργάζεται με τις κατοχώρες με ένα σύστημα το οποίο πραγματικά είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τα, την απόσταση που έχει διανύσει κάθε όχημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ε, ο πρώτος ε, έλεγχος τεχνικής καταλληλότητας θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Στη χώρα μου γίνεται μετά από τέσσερα χρόνια από την αγορά του οχήματος. Εμείς διαπιστώσαμε ότι το να κάνουμε αυτό τον έλεγχο πιο νωρί δεν καταπολεμά την απάτη με τους μετρητές χιλιόμετρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βασίσουμε την πολιτική μας στη συνεργασία την οποία έχουν δημιουργήσει και χτίσει το Βέλιο με τις κατοχώρες. Ας είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει ουσιαστικά να παίρνουμε τις μετρήσεις, να καταγράφουμε τις μετρήσεις του μετρητή και να τις α, πολύ. Ε, ανταλλάσσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Ισμαήλ για την εξαιρετική δουλειά του. Κάτι που θα μας δυσκολέψει εμάς τους και ηγητές γιατί είναι τόσο καλή η έκθεσή του. Ε, το μεγάλο, ε, η αρετή αυτής της έκθεσης είναι ότι ε, ρίχνει φως σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το, η αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά των ε, νέων οχημάτων. 10 εκατομμύρια οχήματα ε, το χρόνο στην Ευρώπη. Ε, τίθενται προβλήματα οικονομικά και ασφάλειας πολύ σημαντικά. Απ' την άλλη μεριά, τα κράτη δεν αντιδρούν, δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα επαρκώς σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τους πολίτες. Πολύ δε περισσότερο που υπάρχουν τρόποι να ελεγχθεί το φαινόμενο. Βλέπουμε το παράδειγμα του Βελίου και των κατοχωρών. Υπάρχει ένα έλεγχο μπορεί να γίνει στο εσωτερικό κάθε χώρας, αλλά όπως λέει και η έκθεση, το 15% των οχημάτων περνούν τα σύνορα και έχω την εντύπωση ότι τα στοιχεία μας υποτιμούν το μέγεθος του προβλήματος, οπότε χρειάζεται να διαθέτουμε και έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό. Αν το σύστημά μας είναι ε, αμυγός εθνικό, ε, θα ενισχυόταν η διασυνοριακή απάτη. Γίνονται τέσσερις προτάσεις στην έκθεση. Πρώτον, η γενίκευση του βαλικού συστήματος, η διασύνδεση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντικό, αυτό είναι το πρώτο. Η πρώτη πρόταση. Δεύτερον, ε, ηλεκτρονικά συστήματα ε, που θα εγκαθίστανται στο όχημα, στο κάθε όχημα. εγώ αναρωτιέμαι πολύ συχνά η απάτη γίνεται από την αρχή της ζωής ενός οχήματος. Δηλαδή ο, ο ίδιος ο ίδιος ο, ο κατασκευαστής ε, είναι το πρώτο θύμα. Δηλαδή παλιά οχήματα πολλούνται σαν να είναι σχεδόν καινούρια. Οπότε και αυτοί και οι κατασκευαστέ ενδεχομένω, η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να ενδιαφερθεί. Γιατί να μην συζητήσουμε και μαζί του. Ε, μετά, νομοθετικό πλαίσιο που να αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο είδο ε, νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι εύκολο να προτείνουμε κάποιο. ε, ε μετά, το blockchain ε, υπάρχει, η αλυσίδα στοιχειών υπάρχει, αλλά είναι πολύ ακριβό, ε, πολύ ακριβός εξοπλισμός. Οπότε ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να δούμε για ποια οχήματα και με ποιο τρόπο διότι μπορεί να δημιουργηθούν και προβλήματα ε, τεχνολογικά και προβλήματα κατανάλωσης ε, καυσίμου. Πάντως πολύ καλή η έκθεση του Ισμαήλ. Ευχαριστώ. vous. κύριος Κράμερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ισμαήλ Ερτούγκ για αυτήν την έκθεση. Πραγματικά είναι εξαιρετική ε, και γι' αυτό είχε και τόσα εγκόμια. Αν λέμε και εγώ και ο Μάρκος ε, Φέρμπερ λέμε πόσο καλά τα πήγε, μήπως κάπου δεν πήγε καλά ο Ισμαήλ, θα αρχίσει να αναρωτιέται. Αλλά ε, Πράγματι, πολύ απλά είναι πολύ καλή η έκθεση. Μπορεί κανεί να ασκήσει κριτικέ. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, πολλά κράτη-μέλη και η Κομισιόν για πολύ καιρό ε, είχαν τεθεί στο πλευρό των απαταιώνων και όχι των τίμιων που είναι και η λύθη της περίπτωσης. Ε, δύο κράτη όμως μας δείχνουν πόσο απλό είναι το πράγμα και δεν έχει βρει μιμητές αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν γίνεται αυτό. Μόνο η απουσία πολιτικής ε, βούλησης ή βούλησης εν γέννη. Και αυτά τα δύο κράτη κάνουν αυτό που πρέπει αλλά υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων και υπάρχουν κράτη που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 δεν έχουν ε, φροντίσει να μην υπάρχει αυτή η παραποίηση και μπορούν να έρθουν αυτά τα αυτοκίνητα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να το εμποδίσουμε. Πράγματι πρέπει να υπάρξει συνδεσιμότητα στην Ευρώπη, θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Πρέπει κάτι να γίνει στην πράξη γιατί προφορικά συμφωνούν όλοι, ούτε έναν επίτροπο ξέρω, ούτε έναν υπουργό μεταφορών δεν ξέρω, ούτε έναν υπουργό δεν ξέρω στα 28 κράτη μέλη που να λέω ότι ναι, πρέπει να στηρίξουμε την απάτη. Φυσικά και όλοι λένε όχι, πρέπει να την καταπολεμήσουμε στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Όμω ε, το πιο απλό θα ήταν ο εκ των υστέρων εξοπλισμό. Ένα ευρώ κοστίζει αυτό το σύστημα για να περιοριστεί η ε, διαδικασία απάτησης, ε, Σχεδόν ψίχουλα θα τα χαρακτήριζα. Και πραγματικά, επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε και διασυνοριακή βάση δεδομένων. Τώρα για το blockchain δεν και τόσο ε, ακριβό βέβαια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση των δεδομένων αλλά δεν σημαίνει ότι ε, θα αλλάξει η κατάσταση παντού. Υπάρχει ε, αποκέντρωση δεν είναι και τόσο ε, κακό ίσως αυτό τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι κάνουμε στην πράξη. Πρέπει και η Κομισιό να πει ότι ναι ε, και εμείς ε, περιμένουμε να υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη. Ε, εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία που θα προτείνουμε βλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για την Κομισιόν να ενεργοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί και να ζητήσει ε, να αναλάβουν δράση τα κράτη-μέλη. Ε, πού υπάρχει το πρόβλημα το γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα. Ότι ναι, στηρίζουμε τους απαταιώνες, ε, θέλουμε αυτοκίνητα φτηνά, παρότι είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να γίνει μια ειλικρινή ανοιχτή συζήτηση. Αυτό θέλουμε εμείς. Θέλω λοιπόν και την υποστήριξή σας να βάλουμε μια ημερομηνία και αυτό θα το κάνουμε εμείς με τη δική μας τροπολογία ε, ώστε να ξεσκεπαστούν αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τους απαταιώνες και να μην την πληρώνουν οι τίμοι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Στρέφομαι αυτή αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, είναι πήγον. Είναι πήγον το ζήτημα. Τι θα μα προτείνετε. Α, κύριε Τελίτσκα, με συγχωρείτε, δεν σα είχα δει. Περιμένετε λίγο από την Κομισιό. Έφτασα αργά γιατί νόμιζα και άλλοι συνάδελφοι θα έπαιρναν το λόγο. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτής της υπόθεσης. Είναι απίστευτο πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο μερικές φορές ρυθμίζουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά διαφεύγουν της προσοχής μας και ταυτόχρονα υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, αφορούν στην εσωτερική αγορά για λόγους οι οποίοι ήδη εντοπίστηκαν και τους είδαμε και εκεί δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ε, πράγματι σκεφτόμαστε κάποιες από τις νομικές ρυθμίσεις οι οποίες υποφέρουν σε επίπεδο εφαρμογής, αλλά στην ουσία χάνουμε εκατομμύρια, έχουμε συγκεκριμένες απειλές στον τομέα της ασφάλειας, έχουμε απειλές στον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω την έκθεση αυτή γιατί ελπίζω ότι θα λειτουργήσει σαν όθηση, σαν κίνητρο, έτσι ώστε η πολιτική εκπροσώπηση γύρω από τα θέματα αυτά σε επίπεδο κρατών μελών να αναβαθμιστεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας από μας εδώ που δεν έχουν επηρεαστεί φίλοι και συγγενείς από τις καταστάσεις εδώ. Ο Πέτερ Γέζεκ, ας πούμε, στην εθνική μου συνιστόσα έχει φύγει από την υπόθεση αυτή. Και ταυτόχρονα, όπως έχουμε πει μέχρι τώρα, υπάρχουν κάποια θετικά συστήματα, διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη. Έχουμε συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τι θα πρέπει να γίνει, αν το σύστημα CarPass είναι επαρκές ή πρέπει να συμπληρωθεί Πάντως περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει επιτέλους δράση. Κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις Νομίζω ότι είναι λογική η έκθεση αυτή, καλύπτει τρεις διαφορετικές επιλογές σε σχέση με τις παραποιήσεις των στοιχείων του αυτοκινήτου και για τις τεχνολογικές λύσεις τώρα και τα μέτρα αποτροπής στα τεχνικά. Νομίζω ότι αν υπάρχει ε, ένα παραθυράκι το οποίο αφήνουν οι κατασκευαστές θα το εκμεταλλευτούν αυτοί οι οποίοι παραποιούν τα στοιχεία. Ε, στη χώρα μου είχε επιχειρηθεί να λειτουργήσει εδώ και δύο χρόνια βέβαια το CarPass αλλά η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγχθει πλήρως. Ο εισηγητής θέλει επίσης να καταστήσει τη συμμετοχή στο νέο σύστημα υποχρεωτική. οι εφαρμογές αυτές βασίζονται σε ένα πλαίσιο νομικό το οποίο μπορεί να είναι διμερές, μπορεί να είναι συνολικό, πρέπει να ελεγχθεί. Και σχετικά με την κυκλοφορία των δεδομένων υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις από ό,τι νομίζω σε χώρες όπως η Γερμανία σαν παράδειγμα τα στοιχεία εντοπισμού ενός οχήματος όπως η πινακίδα κυκλοφορίας καλύπτονται από τις περιορισμούς που θέτει ο νόμος. Είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν κάποια εμπόδια, πρέπει να ξεπεραστούν και η έκθεση αυτή είναι ένα θετικό βήμα και ελπίζω να συνεργαστώ με τους υπεύθυνους. Ευχαριστώ κύριε Τέλιτσκα. θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσατε πόσο κατεπήγον είναι το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια της σε αυτά τα προβλήματα τα οποία θίγουν όλες τις χώρες, θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας και προβλήματα περιβάλλοντος και με οικονομικές απώλειες οι οποίες ε, ε, δεν είναι μόνο εκατομμύρια, μπορεί να μιλήσει κανείς για δις διαφυγόντα έσοδα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το τι σκοπεύει να κάνει στον τομέα αυτό η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλωσορίζουμε την έκθεση ΕΡΤΟΥ. Όπως ε, καθαστήσατε και εσείς σαφές, ε, η απάτη είναι ένα ευρύ φαινόμενο και ε, ένα φαινόμενο το οποίο εμπλέκει πολλές γενικές διευθύνσεις. Τη MOVE, την GROW, ε, για, τον, ε, για την Γενική Διεύθυνση για την Προστασία Καταναλωτών και βέβαια την, ε, έχουμε την πτυχή της απάτης. Εγώ θα σας μιλήσω για το θέμα της ασφάλειας, οδικής ασφάλειας, αλλά έχουμε εδώ συναδέλφους και από την Grow που θα μας μιλήσουν. Ε, να σας κάνω μια σύνοψη του πλαισίου ε, της ε, οδικής ε, συμμόρφωσης, ε, οδικής καταλληλότητας. Έχουμε μια οδηγία για τους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας που εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Θα εφαρμοστεί δηλαδή. Η οδηγία αυτή ο υποχρεώνει σε κάθε έλεγχο να ελέγχεται και η ακαιρεότητα του μετρητή χιλιόμετρων. Και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ε, διαθέσιμα και για τον επόμενο έλεγχο. Επίσης, ε, οποιαδήποτε αλλίωση του μετρητή θα πρέπει να αποτελεί αδίκημα για όλα τα κράτη-μέλη από το Μάιο του 2018 και μετά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι βέβαια μια οριστική και ολοκληρωμένη λύση, αλλά από φέτος θα έχουμε ήδη δεδομένα και την υποχρέωση να ε, να, είναι, να αποτελεί αδίκημα η αλλίωση των μετρήσεων. Τώρα, λέτε ότι η, έκθεση μάλλον λέει ότι η Κομισιόν δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της ε, να θεσπίσει διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο όμως η υποχρέωση της Κομισιόν ήταν μόνο μια μελέτη βιωσιμότητας. Η πρόταση για ένα σύστημα διασυνορικής ανταλλαγής πληροφοριών ε, θα ήταν μια καινούρια πρόταση που ξεφεύγει από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε καθορίσει. Τώρα βέβαια, συμφωνούμε με σας ότι είναι πολύ σημαντική η διασυνορική ανταλλαγή πληροφοριών και θα διευκόλυνε σαφέστατα σε ένα μεγάλο ή σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων την καταπολέμηση των, της απάτης για τους μετρητές χιλιόμετρων. Και θα ήταν σημαντικό να ανταλλάσσουμε και άλλα στοιχεία, όχι μόνο τα στοιχεία των μετρητών. Η, αυτή η ανταλλαγή θα ήταν πιο ευρεία λοιπόν και θα ωφελούσε και τους χρήστες και τις αρχές. Τα, το, το νομοθετικό πλαίσιο για την τεχνική, για τεχνική καταλληλότητα περιλαμβάνει μέτρα για τις αρχές και αυτές οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται θα τη χάνουν διαχείρισης από τις ίδιες κρατικές αρχές. Συνεπώς η ανταλλαγή θα γίνεται μεταξύ κρατικών αρχών. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή λύση στο πρόβλημα. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών χωρίς ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Eucaris, το σύστημα πληροφοριών, αυτοκινήτων και αδειών οδηγηση, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο τη τεχνολογία και να μην εμπλέκονται τα κράτη-μέλη. Τώρα, για τα θέματα προστασίας του καταναλωτή. Αναγνωρίζουμε πως είναι σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία, όπως είπα, θα διαχειριζόνται οι ίδιες οι εθνικές αρχές. Εξετάζουμε το πώ αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα στο πλαίσιο ελέγχου τεχνικής καταλληλότητας ή μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Θα δούμε. Επίσης, η έκθεση προτείνει ε, ο πρώτος έλεγχος τεχνικής καταλληλότητας να περάσει από τον τέταρτο στον τρίτο χρόνο ζωής του οχήματος. Δεν συμφωνούμε με την έκθεση. Γιατί, Γιατί στην πράξη μην ξεχνάμε ότι οι έλεγχοι τεχνικής καταλληλότητας έχουν ως στόχο να ε, ελέγχεται το κατά πόσον το όχημα τηρείται σε κατάσταση ε, τεχνικής και οδικής ασφάλειας. Ε, οι μετρητές χιλιόμετρων είναι ένα κομμάτι από τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, αλλά ένα μικρό κομμάτι θα πρέπει να εξετάσει, για παράδειγμα αν τα ελαστικά βρίσκονται σε σωστή, κατάσταση, τα φώτα κλπ. Και ένα αυτοκίνητο που περνάει το τεστ ε, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση ακόμα και αν έχει αλλοιωθεί, ο, έχει παραποιηθεί ο μετρητής. Ε, αλλά ο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα, οι μετρητές είναι θέμα καταναλωτή, προστασία καταναλωτή, ενώ ο τεχνικός έλεγχος είναι θέμα ασφάλειας, οδικής ασφάλειας. Ε, το Βέλγιο και η Ολλανδία έχουν ένα σύστημα, η Σλοβακία ε, ε, προετοιμάζει το δικό της σύστημα και τα κράτη-μέλη μπορούν να προσθέσουν καινούριου ελέγχους ε, για να αντιμετωπίσουν το θέμα της απάτης με τους μετερτές Πριν από ένα χρόνο ξανά είναι αυτή η συζήτηση και σας ακούσα πολύ προσεκτικά. Εν τω μεταξύ εμείς τι κάναμε, κάναμε ένα-δύο πραγματάκια. Τι κάναμε, ε, προσθέσαμε ε, το θέμα του προσθέσαμε τον έλεγχο των μετρητών στους ε, τακτικούς ε, ελέγχους κταίου που γίνονται. Ε, επίσης, ε, αποφασίσαμε να προωθήσουμε τις καλές βέλτιστες εθνικές πρακτικές και το κάνουμε ήδη, προσπαθούμε δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αντιγράψουν τα παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συμπληρώσουμε το ε, νομικό πλαίσιο για τους έλεγχους τεχνικής καταλληλότητας προσθέτοντας τον έλεγχο των μετρητών. Νομίζουμε ότι προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Το κοινοβούλιο μας ενέκρινε ένα πλειοτικό πρόγραμμα για την ε, πειραματική ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα μετρητών ε, χιλιόμετρων και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα για να κάνουμε μια λεπτομερή ανάλυση και ενδεχομένως και μια ε, ανάλυση αντικτύπου και μια νομοθετική πρόταση ενδεχομένως ε, για την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων. Τέλος, προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, επεξεργαζόμαστε μια, ένα καινούριο πλαίσιο πολιτικής για την οδική ασφάλεια για την ερχόμενη δεκαετία ως τμήμα του τρίτου πακέτου κινητικότητας ε, που θα δημοσιευθεί την Άνοιξη θα αναλύσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία και θα διαπιστώσουμε πού χρειάζονται τροποποίησεις. Η, η τεχνική ειδική καταλληλότητα ίσως είναι πιθανότατα θα είναι ένα από τα θέματα για τα οποία θα χρειαστούν ε, τροποποιήσεις. Ε, κάλυψα, λοιπόν το θέμα της τεχνικής καταλληλότητας, όμως οι συνάλφοι από την Γενική Διεύθυνση ε, Grow μπορεί να θέλουν να μιλήσουν για το θέμα της έγκρισης τύπου. Πρόεδρος, Ευχαριστώ για, την, ε, για τα σχόλιά σας, αλλά πραγματικά μου δημιουργεί σημαντικές ε, αμφιβολίες και δισταγμούς η ε, τοποθέτησή σας. Λέτε δεν έχουμε υποχρεώσεις γιατί περιμένουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση από τη συνθήκη για την οδική ασφάλεια, για θέματα κατα... Ε, ε, περιβάλλοντος και δικαιωμάτων καταναλωτή. Και εσείς τι μας λέτε, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια, ας αφήσουμε τα κράτη-μέλη. Τι περιμένουμε. Να γίνει ένα σκάνδαλο όπως το Dieselgate. Να έρθουν να έρθει κάποια άλλη χώρα να μας πει ότι, όπως έγινε με το Dieselgate, ότι τα αυτοκίνητα μας έχουν πρόβλημα. Δεν είναι δυνατό να μας λέτε ε, ότι αρκεί τα κράτη-μέλη ε, να καταστήσουν ε, ποινικό αδίκημα την παραποίηση. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Μετά λέτε από το Μάη θα ελέγχονται οι μετρητές στους ελέγχους κτεο χωρίς όμως περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Κομισιόν είχε πει ότι θα, το θέμα αυτό θα το καταστήσει προτεραιότητά της. Έχει δεν το κάνει. Πρέπει να σας πω ότι οι φιλοδοξίες σας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Εμείς από την άλλη μεριά σας λέω ότι θα το θέσουμε πραγματική προτεραιότητα. Γιατί οι πολίτες μας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η απάτη. Συνεπώς, παρακαλώ πολύ, σας ζητώ για άλλη μια φορά να μας προτείνετε συγκεκριμένες δράσεις. Θα δώσω την γενική, ε, το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Grow, να δούμε τι καινούργια στοιχεία μπορεί να μας δώσει και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Άρτουκ να πάρει το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγκεντρωθώ στα τεχνικά χαρακτηριστικά της έκθεσης. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι, έχουμε προχωρήσει προς την κατάφυση αυτή ε, σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου 2.17 11.51. Είναι ήδη ενισχύ από τον προηγούμενο Ιούλιο η νομοθετική αυτή ρύθμιση απαιτεί τον κατασκευαστή να έχει μέτρα αποτρεπτικά για παρεμβάσεις στον χιλιομετρητή. Η μέθοδος αυτή εγκρίνεται και από την αρχή έγκρισης τύπου. Υπάρχει ξεχωριστός ρόλος των δύο αυτών επιπέδων. Συνεπώς λοιπόν το πρώτο σας αίτημα το λαμβάνουμε υπόψη θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή. Στις, 18 Φεβρουαρίου έχουμε μια, στις 8 Φεβρουαρίου έχουμε μια συνάντηση με τις αρχές έγκρισης τύπου και θα δούμε πώς εφαρμόζεται η ρύθμιση. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ένα δεύτερο ε, επίπεδο σχετικά με ε, τα συστήματα καταγραφής της κατανάλωσης. Information measure. Ναι, ναι. Ταυτόχρονα ε, προσπαθούμε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια του καθεστώτος των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα γρήγορα και εδώ. Ένα τελευταίο στοιχείο να προσθέσω ότι θα εξετάσουμε το δεύτερο τμήμα των συστάσεών σας που ζητούν μέτρα και σε επίπεδο λογιστικό και σε επίπεδο λογισμικό. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις ε, με το Κοινό Κέντρο Έρευνας και ελπίζουμε να έχουμε κάποια στοιχεία ε, σε υστερότερη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο ένα λεπτό κύριε Χέρτογκ στον Βαντερκάμπ και μετά θα πάρετε εσείς το λόγο για δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Εμείς εργαζόμαστε χρόνια με την υπόθεση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με εκατοντάδες θέματα, αλλά με το θέμα αυτό το οποίο άπτεται άμεσα των πολιτών, φοβάμαι ότι είναι πολύ επιφυλακτική. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε και θα πρέπει η Επιτροπή να ενθαρρύνει και αυτή ε, τα κράτη-μέλη. Τι θα πει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ανεπαρκές, είναι ασθενές σαν μέτρο. Και αναφέρομαι όχι σε θέματα έγκρισης τύπου, σε μεταχειρισμένα οχήματα. Τα μεταχειρισμένα οχήματα είναι αυτά τα οποία υφίστανται τις απάτες. θα πρέπει επιτέλους το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί. Έχουμε ευθύνε ε, στους εκλογείς μα. συζητάμε τα θέματα αυτά μαζί τους, όχι μόνο το Brexit όμως, έχουμε εδώ ε, θέματα πολύ σημαντικών απατών. Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Βαντερκάμπ, ο, Χερ, ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ του ε, συναδέλφου ε, και την Κομισιόν. Πριν έρθω στην Κομισιόν, ε, σε ό,τι αφορά τα φορτικά, επειδή μου κάνατε μια ερώτηση προηγουμένω. Αρχικά και εμείς τα σκεφτήκαμε και το συστήσαμε και με τους εμπειρογνώμονες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αντίστοιχη απάτη στα φορτηγά όπως τα οχήματα με κινητήρα γιατί υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής ε, των διαδρομών και ο ταχογράφος ταυτόχρονα οπότε καταγράφεται παράλληλα και από τα δύο συστήματα ε, ο αριθμός των διανυθέντων ε, χιλιόμετρων οπότε θεωρούμε και το λένε και οι εμπειρογνώμονες αυτό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραποίησης των στοιχείων. Τώρα, έρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα μας είπαν και διαπιστώνω ότι παρά τις πολλές επαφές και συζητήσεις που έχουμε εδώ και ένα μισό χρόνο με την Κομισιόν και τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, πραγματικά δεν φεύγει από το μυαλό μου και δεν φεύγει αυτή η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ επιφυλακτική και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Είναι πολύ επιφυλακτική για θέματα ε, που ε, τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να ε, τους, να απαιτήσουμε από αυτά να προβούν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Δηλαδή, ο κόσμος ε, πολύ σωστά πιστεύω ε, καταλαβαίνει και νιώθει ότι δεν τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη και ότι αυτά τα θεωρεί ασήμαντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε όμως για τους ε, καταναλωτές. Και πραγματικά πρέπει να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν αυτοί οι τύποι στις Βρυξέλλες εκεί αφιψηλού. Με τη βοήθειά σας αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το πούμε ορίστε να τι έχουμε κάνει με την ε, παραποίηση, με την απάτη, με τι έχουμε καταφέρει τέλος πάντων για εσάς. Πρέπει κάποια στιγμή να το πετύχουμε αυτό δεν θα υπάρχουν επιχειρήματα πλέον για να το υποστηρίξουμε. Είναι ε, ένα παράδειγμα αυτό για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και πράγματι ε, είναι θέμα νομοθεσίας. Έχουμε και την περσινή νομοθεσία και όλα αυτά. Αλλά σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου. Έχει να κάνει με την έγκριση, με την ταξινόμηση, την πρώτη ταξινόμηση. Εμείς λέμε τι γίνεται μετά ε, με τα μεταχειρισμένα οχήματα. Αυτό μας απασχολεί. Θέλουμε λοιπόν να εισαχθεί ένας θεσπισμός από την πρώτη αξινόμηση μέχρι τον πρώτο ε, τεχνικό έλεγχο. Τέσσερα χρόνια είναι ε, το διάστημα αυτό. Σε αυτή την τετραετία δεν θέλουμε να υπάρξει δυνατότητα παραποίησης. Δεν προβλέπεται κάτι από την νομοθεσία, την υφιστάμενη, για αυτά τα τέσσερα χρόνια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ευρωπαϊκή ανταλλαγή με τα μεταχειρισμένα Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα κράτη-μέλη. Πρέπει να λάβουν τα, ε, τις ευθύνες τους. Δεν ξέρω αν θα είναι το γιουκάρις ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Δεν είναι το αποφασιστικό για μας ποιο σύστημα θα εφαρμοστεί. Αυτό που κατέσσε σαφές νομίζω εδώ είναι ότι υπάρχει συνένεση ευρεία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, ο κύριος Κράμερ, ένα λεπτό, τι θέλετε. Πολύ πιο σύντομο. Τα έχουμε συζητήσει. Για την προστασία των καταναλωτών, γιατί δεν μίλησε κανένας. Αυτή είναι τα θύματα καθημερινά της απάτης αυτής. Έχουν άλλη άποψη από εσάς, τις άλλες υπηρεσίες που μιλήσατε. Γιατί δεν μίλησαν. Ευχαριστώ κύριε Κρέμερ. Ε, η, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Φεβρουαρίου. Και θα σας πληροφορήσω ότι η έκθεση αυτή θα προωθηθεί στο Κοινοβούλιο και θα ζητήσουμε από την Κομισιόν ένα σαφή οδικό χάρτη. Και κυρίως ένα οδικό χάρτη που θα αποτελεί χάρτη δράσης. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια ενώ η απάτη εκτινάσεται προσβάλλοντας τα, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών και δημιουργώντας σημαντικές οικονομικές ζημίες. Ε, πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να μην προστατεύει αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προστατεύει αυτά που αγοράζουν οι καταναλωτές θέλουμε να σπρώξουμε την Κομισιό να αναλάβει δράση σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να βρεθούμε αύριο μεθαύριο ε, να βρεθούμε σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που βρεθήκαμε στο σκάνδαλο του Dieselgate. Διακοπή διάλειμμα για 10 λεπτά και μετά θα υποδεχθούμε την Βουλγαρική Προεδρία. Ευχαριστώ.

Ευχαριστώ.

Mes chers collègues, nous Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναξεκινάμε ε, με την ε, μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε εδώ τον Βούλγαρο Πρόεδρο Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Μοσκόφσκι. για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Μεγάλη χαρά Μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε σήμερα. Puisque la Bulgarie a pris la présidence le 1er janvier avec beaucoup d'ambition. Ξεκινάμε αυτή τη χρονιά με μεγάλη φιλοδοξία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέρχεται μια δύσκολη περίοδο αλλά μας διακατέχει ενθουσιασμός ε, θέλουμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Μέσα στις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας έχετε θέματα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας, ιδιαίτερα στους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Βουλγαρική Προεδρία και να σας δώσω το λόγο ευχαριστώντας σας που είστε μαζί μας σήμερα. Να επανέλθετε μάλιστα όποτε το επιθυμείτε έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τον οδικό σας χάρτη για τους επόμενους έξι μήνες. Σας δίνω το λόγο για 20 περίπου λεπτά και μετά θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι συγκινητική στιγμή για μας. Και για μένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή που θα σας παρουσιάσω σήμερα τις ε, προτεραιότητες μας για θέματα μεταφορών, θέματα που θα συζητηθούν στο επόμενο εξάμεινο. Η Βουλγαρία έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να συμμετάσχει δραστήρια στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας, καθώς επίσης και τη δική σας ευθύνη, διότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που να κοιτούν το μέλλον με βάση την αρχή της δεκτικότητας και της διαφάνειας. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρική Προεδρία θα προωθήσει τη συνένεση, την ανταγωνιστικότητα και την σύνοχη σε όλους τους τομείς του κλάδου των μεταφορών. Συμπεριλαμβανομένης και της ε, εμβάθυνσης της συνεργασίας έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να ε, εκτεθούν και να ε, υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές αρχές. Χάρη στην ε, θέση της στη Βαλκανική Χερσόνησο, η Βουλγαρία πάντοτε έπαιζε το ρόλο, ανάμεσα στην γέφυρα, ε, το ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων ε, και αγαθών. Και αυτόν τον ρόλο συνεχίζουμε να παίζουμε, ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλη την Ευρώπη. Ο κλάδος των μεταφορών μπορεί να ε, βοηθήσει την οικονομική για της Ευρώπης, αλλά και την περιφερειακή συνοχή και την ευημερία των πολιτών μας. Η Βουλγαρική Προεδρία θέλει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τομέα, εργαζόμενοι κυρίως κατά προτεραιότητα επί πρωτοβουλειών που ε, προέρχονται από το πρώτο και το δεύτερο πακέτο κινητικότητας και, για τις, και επί των νομοθετικών πράξεων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική των Εθέρων. Αναλαμβάνουμε την ε, Προεδρία σε μια στιγμή κλειδί για τη διαπραγμάτευση του πρώτου πακέτου κινητικότητας η ολοκλήρωση της εργασίας ε, επί των διαπραγματεύσεων που έχει αναλάβει το τρίο των ε, Προεδριών θα μας οδηγήσει σε μια Ευρώπη πιο ευημερούσα. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες για το ε, θέμα που έχει σχέση με την πρόσβαση στις αγοράες και την πρόσβαση στο επάγγελμα. Επίσης, τις εργασίες σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις οδηγών τα ενοικιασμένα οχήματα και την διαλειτουργικότητα των τηλεδιοδίων. Οι κοινωνικές πτυχές ε, και η απόσπαση των εργαζομένων έχουν καταστεί πολιτικά ως ευαίσθητα θέματα στην Ευρώπη. Η συζήτηση ελπίζω ότι θα είναι επικοδομητική και σε βάθος για αυτά τα δύο θέματα. Οι νομοθετικές προτάσεις του πρώτου πακέτου κινητικότητας θα πρέπει να βασιστούν σε δίκες και ισορροπημένες προτάσεις. Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί να προστατευτούν και να προσφέρουν την υπηρεσίες τους ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι σαφείς κανόνες και οι καλή έλεγχη είναι πάρα πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προστασία ε, του ανταγωνισμού. Η χρήση νέων τεχνολογιών θα μας επιτρέψει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Ευρώπη άλλωστε θα μας επιτρέψει ε, να κάνουμε την αγορά πιο ανταγωνιστική η υιοθέτηση μιας γενικής προσέγγισης για αυτό το θέμα θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα, μια πρόοδο την οποία ελπίζω ότι θα πετύχουμε προκειμένου να θέσουμε σωστές βάσεις ε, για τις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα στην επόμενη Προεδρία. Μετά, οι ε, συνδυασμένες μεταφορές ε, η Προεδρία της, η Βουλγαρική Προεδρία ήδη ξεκίνησε τις εργασίες σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους κοινού κανόνες συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων την αναδιατύπωση της οδηγίας η οποία υιοθετήθηκε πριν από 25 χρόνια και δεν έχει μεταγραφεί με ίδιο ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη κάτι που περιορίζει το δυναμικό της. Η μετάβαση από τις χερσαίες μεταφορές ε, μεγάλης, ε, ε, μεγάλων αποστάσεων ε, στην μεταφορά δια της πλωτής οδού ή με τους σιδηροδρόμους θα οδηγεί στη βελτίωση της χρήσης των οδικών μεταφορών και η καλή εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα βοηθήσει τον κλάδο ο οποίος θα πρέπει να έχει κίνητρα για να κάνει αυτή τη μεταφορά τη μετάβαση, συγγνώμη. Η αναθεωρημένη οδηγία θα συνεισφέρει στην δημιουργία περισσότερων συνδέσεων με διάφορα μέσα μεταφοράς που θα προσθεθούν στους, στις συνδέσεις που ήδη υπάρχουν και επίσης θα οδηγήσει στην δημιουργία καινούριων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη. Η, ε, το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην συνάντηση ψηλού επίπεδου των Υπουργών Μεταφορών που θα λάβει η χώρα στις 19 και 20 Μαρτίου στην Σόφια. Οι δυνατότητες ανταλλαγής εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας απαιτούν ε, την ε, ενίσχυση των μεταφορών μέσω του Δούναμπη και της Μαύρης ε, Θάλασσας, καθώς επίσης και την ε, χρήση των διευρωπαϊκών δικτύων. Η, συνεργασία με τις χώρες αυτών των περιοχών είναι πάρα πολύ σημαντική για να βελτιωθούν οι υποδομές. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να συντονίσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας και επίσης να εξασφαλίσουμε και χρηματοδότηση για ένα ασφαλές, ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκτυο μεταφορών στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασύνδεσης στην Ευρώπη, ε, καθώς επίσης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να βελτιώσουμε τη συνεργασία στην περιοχή των Βαλκανίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εναέριες μεταφορές. Ε, έχουμε τον κανονισμό για την προστασία του, ε, του ανταγωνισμού στον ε, τομέα των εναέριων μεταφορών και αυτό είναι προτεραιότητά μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις μεταφορές από πολιτικές αλλίωση του ανταγωνισμού τρίτων χωρών ε, και αναμένουμε ο, ο κανονισμός αυτός να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να δώσει στους πολίτες περισσότερες επιλογές μειώνοντας τις τιμές μακροπρόθεσμα χωρίς αυτό να μειώσει την διασύνδεση των περιφερειακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την διασύνδεση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. αν δεν αντιδράσουμε στις ε, ε πρακτικές στρέβλος του ανταγωνισμού μπορεί να οδηγηθούμε σε δεσπόζουσες θέσεις ή και σε μονοπόλια στην ε, αγορά αυτή. Κάτι που θα περιόριζε πάρα πολύ τις επιλογές των ε, καταναλωτών μας, θα μείνουν την ποιότητα και θα αύξαναν τις τιμές. Αυτή η νομοθετική πρόταση θεωρείται από τα κράτη-μέλη ως αντιφατική. Αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η μοίρα κάθε νομοθετικής πρότασης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή θέστηση των κρατών μελών. Θα πρέπει ο κανονισμός να συνάδει με τις διασύνδεσμας μα υποχρεώσεις. θα πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσει με τρίτες χώρες προκειμένου να συνάψουμε διμερείς σχέσεις που να λαμβάνουν υπόψη το δικό μας κεκτημένο. Αυτές οι συμφωνίες θα εγγυώνται τον υγιή ανταγωνισμό, την ίση μεταχείριση, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η Βουλγαρική Προεδρία θα συνεχίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά θα καλωσορίσουμε και οποιαδήποτε καινούρια πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η Βουλγαρική Προεδρία θα εργαστεί επί μιας καινούριας ε, ε, οδηγίας ε, για λιμενικές εγκαταστάσεις αποθήκευση και επεξεργασίας λιμάτων από τα πλοία. Αυτή η οδηγία θα οδηγήσει σε, βελτιστη, σε βελτιωμένη προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος και θα μειώσει επίσης και τα, το διοικητικό άχθος των επιχειρήσεων. Η πρόταση οδηγίας ε, σχετική με την ευρωπαϊκή μονοπευθυντική θηρίδα θα υποβληθεί το 2018 για πρώτη φορά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί θα διευκολύνει ε, τις ε, επιχειρήσεις ε, που ασχολούνται με το εμπόριο μέσω θαλάσσης. Εμείς θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επί αυτής τη πρότασης μόλις μας την παρουσιάσει η Κομισιόν. Η Κομισιόν επίσης θα υποβάλει πρόταση αναθεώρησης οδηγίας για το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης ε, των επαγγελματών τη θάλασσα, καθώς επίσης και την πρότασή τη για την οδηγία περί αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων του και των διπλωμάτων τους. Ε, επίσης θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες σε ό,τι αφορά την σύσταση του Συμβουλίου για τις απαιτήσει ε, που βαρύνουν τα μικρά σκάφη. Η Βουλγαρική Προεδρία ε, θα διοργανώσει την ετήσια, ε, ένα ετήσιο συνέδριο, μια, μια ε, ημερίδα στο Μπουργκάς από τις 30 Ιουνίου μέχρι την, 30 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου ε, για τα θέματα της γαλάζιας ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τις ιδεοδρομικές μεταφορές, θέλουμε να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, επιβατών, κάτι που θα οδηγήσει σε βελτίωση της, των υπηρεσιών που παρέχονται. Προβλέπουμε και εδώ συνέδριο για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού το μέλλον του, ε, τη σύνδεση, ε, τις και την ε, θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο Μεταφορών ε, θα συνεδριάσει 7 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω τελειώνοντας ότι θα χρειαστούμε τη συνεργασία σας και την υποστήριξή σας για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Οι πολίτες μας περιμένουν από μας απαντήσεις σε ε, θέματα τα οποία χρονίζουν. Θέλουμε να βασιστούμε στη δική σας συνεργασία, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η περίοδος είναι ε, ρευστή. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και ακούει τις ανησυχίες των πολιτών της. Τα αποτελέσματα των σημερινών αποφάσεων θα πρέπει να επηρεάζουν αμέσως αύριο τις ζωές των πολιτών μας. Το 57% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύει στην Ευρώπη εμπιστεύεται την Ευρώπη. Πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στις χώρες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι το, μέρος, το πιο καλό μέρος για να ζει κάποιος στον κόσμο σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και τι περιμένουν από εμά οι πολίτε μα, πιο συντονισμένε δράσει, λύσει στα προβλήματά του. Απαιτούν μια Ευρώπη πιο ε, δίκαιη, μια Ευρώπη που να δημιουργεί ανάπτυξη. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το σύνθημα της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας είναι ε, η Ένωση μας κάνει πιο δυνατούς. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Monsieur. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρέμβαση αυτή. Ήσασταν πολύ συγκεκριμένος. Πώς θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις ε, για την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί σήμερα κανένας συμπολίτης μας δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τις συγκοινωνίες, χωρίς μεταφορές. Η κινητικότητα ήταν ένα εργαλείο που επέτρεψε στους πολίτες να ανακαλύψουν διαφορετικούς τόπους, διαφορετικά μέρη, αλλά αλλάζει και την καθημερινότητά τους, πώς πάνε στη δουλειά τους, πώς πάνε στο σχολείο. για την ψυχαγωγία του, την αναψυχή του, ε, να πάνε στο κέντρο τη πόλη να ψωνίσουν κτλ. κτλ. Μεταφορές, συγκοινωνία σημαίνει καθημερινότητα. Πολίτε σήμερα χάνουν πολύ χρόνο ε, στα μέσα μεταφοράς, αλλά προσβασιμότητα, άνεση έχουν βελτιωθεί. Υπάρχουν προκλήσεις σίγουρα, κλιματικές, περιβαλλοντικές, αλλά και προκλήσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Κύριε Υπουργέ, πολύ σωστά μας ζητήσατε να στραφούμε προς το μέλλον. Και είπατε ποιο είναι το σλόγγαν της ε, Προεδρίας σας η ισχύσει εν τη ενώση. Πράγματι, αυτό ισχύει. Και υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ τη ονομαθία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Για τα κοινωνικά θέματα επίση, ναι, πρέπει να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και να σημειώσουμε πρόοδο και στο κοινωνικό επίπεδο. Είπατε ότι έχετε τη διάθεση και τη βούληση να βοηθήσετε αυτό πολύ σημαντικό εργαλείο της απασχόλησης να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την ανάκαψη. Μπορείτε να βασίζεστε στην Επιτροπή Μεταφορών, στην καλή μας θέληση, στην αποφασιστικότητά μας. Γιατί είμαστε μια ομάδα. Και στόχος μας είναι να πετύχουμε τους ίδιους στόχους. Θα ξεκινήσω τώρα αυτή αμέσω τη συζήτηση, δίνοντα καταρχά πρώτα τον λόγο στου συντονιστέ και έπειτα σε όποιον άλλο συνάδελφο το επιθυμεί. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Βιμ Βαντενκάμπ, συντονιστής από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, κύριε Βαντενκάμπ. Θα έχετε το λόγο πρώτος. Ε, θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Τρία λεπτά θα έχουν στη διάθεσή τους οι συντονιστές και οι υπόλοιποι δύο. Θα είμαι πολύ αυστηρή, με ξέρετε. Κύριε Βαντενκάμπ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Συγκοινωνιών μεταφορών μάλλον της Βουλγαρίας. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την πρώτη Βουλγαρική Προεδρία. Είναι ιστορικό το συμβάν. Γνωρίζουμε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε τις εντάσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και αυτά τα οποία μας είπε ο Υπουργός είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί θα επιτρέψουν να υπάρξουν σωστές συνδέσεις ανάμεσα σε όλες αυτές τις χώρες. Να πω επίσης ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να θέλουν πράξεις συγκεκριμένες από πλευράς μας και όχι να μένουμε σε επίπεδο αρχών και λόγων. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν με αυτό τρόπο αυτό το οποίο κάνουμε. Το Σεπτέμβριο του 2017 ήμουν στη Σόφια κύριε Υπουργέ ε, συναντήσαμε και την Επιτροπή Μεταφορών του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Είδαμε ότι η Βουλγαρία είναι μια σημαντική χώρα, ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές. Και όταν ξεκινήσετε τη δουλειά στο Mobility 1, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και μεγάλη πρόκληση για όλους, ιδιαίτερα για να υπάρξει κοινή θέση στο Συμβούλιο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θέματα της απόσπασης των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Mobility 1 και θέλουμε να προχωρήσουμε και στο Mobility 2. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αναλάβουμε υποχρεώσεις περισσότερες από όσες μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 19. Αναφερθήκατε στο ότι η Βουλγαρία είναι πράγματι σημαντική χώρα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν αρκετά θέματα και προβλήματα στη σύνδεση και της δικής σας χώρας με άλλες χώρες και μεταξύ των άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας πήγαμε στον λιμένα του Μπουργάς και είδαμε τη σημασία που έχουν και οι θαλάσσιες μεταφορές. Σας άκουσα να μιλάτε και για τον Δούναβη ο Δούναβης ε, είναι μια σημαντική συνδετήρια οδός στα πλαίσια των TNT. Είναι μια μόνιμη πρόκληση και ενδιαφέρομαι ε, πώς συνεργάζεστε με τη Ρουμανία στο συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Βαντερκάμπ, δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κουρούμπασεφ. Είδατε, σας το είπα και με προφορά. Πράγματι, πολύ ενδιαφέρουσα η προφορά σας. Αγαπητέ Υπουργέ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας καλωσορίζω εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε στην Βουλγαρία και το νησί που επισκεφθήκαμε λέγεται Αγία Αναστασία, κοντά στο Μπουργκάς. Έμαθα χθε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν θα υποστηρίξει τα δίκτυα ε, μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια. Και εσείς εκπροσωπείτε, ε, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Βουλγαρία. Θέλετε να επιμείνετε τι θα κάνετε για την ανάπτυξη των ε, περιφερειακών μεταφορών. Είναι μια βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής σας, αλλά ε, στον τομέα των μεταφορών ειδικά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μένει να γίνουν. Η διαδικασία οι διαδικασίες ε, που θα οδηγήσουν στην ε, ένταξη των χωρών της περιοχής θα διευκολυνθούν από την ανάπτυξη των μεταφορών. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα βελτιώσετε τη διασύνδεση ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αδριατική Θάλασσα. και η δουλειά την οποία έχουμε μπροστά μας στον τομέα της απόσπασης των εργαζομένων είναι τρομακτικά δύσκολη. Βλέπω ότι υπάρχουν περισσότερες εθνικές διαφορές μερικές φορές, πιο ισχυρές από ότι ε, διαφορές ανάμεσα σε χώρες και κάτι τέτοιο θα καταστήσει τη δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο πολύ δύσκολη. Ελπίζω να μπορέσετε να εξισορροπήσετε τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών μελών λοιπόν και ελπίζω επίσης ότι θα καταφέρετε να μας οδηγήσετε σε μια συνενετική θέση. Ο κύριος Καμπ αναφέρθηκε επίσης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να μας δώσετε για την ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή αυτή στα πλαίσια της συνεργασίας ε, με χώρες όπως η Αρμενία και η Γεωργία. Υπάρχει προοπτική σύνδεσης πέραν της Τουρκίας ε, με το Ιράν και την Μέση Ανατολή. Ξέρω ότι υπάρχουν επίσης και αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται στις, για την πρωτοβουλία ε, γύρω από τον Δούναβη. Ποια είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Με χαρά σας συναντώ κύριε Υπουργέ και θέλω να ευχηθώ κάθε καλό και κάθε επιτυχία στην Προεδρία της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι μπορείτε πράγματι να πετύχετε. Είχαμε συναντηθεί τον Νοέμβριο στη Σόφια, είχαμε την τύχη να συναντήσουμε τους εκπροσώπους όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της κυβέρνησης και χαίρομαι που και η αντιπολίτευση της χώρας είπε ότι θα υπάρξει εξάμεινη ανακοχή ε, έτσι ώστε να μπορέσει ανεμπόδεστα η κυβέρνηση να καλύψει και τις ανάγκες της ε, Προεδρίας. Το θέμα λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι του Mobility, το Mobility 1. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να πετύχετε τους στόχους, αλλά εν περιπτώσει η προσπάθεια που θα γίνει ε, νομίζω ότι θα είναι ικανοποιητική. Πώς μπορείτε λοιπόν να δράσετε έτσι ώστε στον τομέα των μεταφορών να υπάρξει μια ενιαιοποίηση της αγοράς σας στην περιοχή σας Ξέρουμε ότι η περίπτωση του Καμποτάζ σαν παράδειγμα και η περίπτωση της εσωτερικής αγοράς είναι δύο στοιχεία που συνδυάζονται μεν, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Σαν παράδειγμα η απόσπαση των εργαζομένων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή, αλλά θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον διοικητικό κόστος για τον έλεγχο του καμποτάζ έτσι ώστε να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων. Και για το Mobility 2, εγώ έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος για τις τροπολογίες σχετικά με τον κανονισμό για τα λοφορία διεθνών μεταφορών. Η κατάσταση δεν έχει μετακινηθεί ιδιαίτερα, οι εξελίξεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, οπότε τι γίνεται με τις επιβατικές οδικές μεταφορές μέσω λεωφορείων. Και μία τρίτη ερώτηση αφορά το επόμενο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο Μεταφορών θα οργανωθεί τον μήνα Ιούνιο. Θα ήθελα να μάθω ποια θα είναι η αντίδραση της Προεδρίας σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τέλιτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι καλή τύχη. Έχετε το πλεονέκτημα αλλά και την πρόκληση να ε, ακολουθείτε μια πετυχημένη προεδρία. Σας, ε, σας εύχομαι να είστε εξίσου πετυχημένοι κι εσείς. Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να φύγω σύντομα, ε, αλλά θα ήθελα να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Κάτι που είπατε σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε αυτό το θέμα ως στοιχείο της συζήτησης. Αν μπορούσατε μάλιστα να αναλύσετε, να αξιολογήσετε και να μετρήσετε τον αντίκτυπο Τη χρηματοδότηση που είχαμε μέχρι τώρα και να βγάλετε και κάποια συμπεράσματα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δεύτερον, μιλήσατε για τον ανταγωνισμό στις ενέργειε μεταφορές. Προφανώς ε, είμαστε σε ένα πρώτο στάδιο. Πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία μονοπωλίων και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οπότε μιλήσατε για την προστασία των καταναλωτών, αλλά μήπως μπορούσαμε να δούμε και τη δεύτερη πτυχή του θέματος, που είναι πια ότι για να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μας κάνουν ανταγωνιστικούς, όχι μόνο την προστασία του καταναλωτή. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε πολλές λεπτομέρειες για όλα αυτά τα θέματα που σχολιάσατε. Ούτε και εγώ θα σας ζητήσω λεπτομέρειες βέβαια. Θα έχουμε χρόνο ε, να τα δούμε αυτά με τους συναδέλφους σας ε, στο μέλλον. Όμως, ποιος είναι ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η Βουλγαρική Προεδρία σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητα 1, το πακέτο 2 και στο μέλλον και για το θέμα των ενέργειων μεταφορών. Καλό είναι να τα ακούσουμε και από το στόμα σας. Σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητα, νομίζω ότι ο βασικό δικός μας στόχο είναι ε, να λειτουργεί μια εσωτερική αγορά ε, χωρίς ε, στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και με βάση αυτό το στόχο θα κρίνουμε την πρόοδο. Σίγουρα χρειαζόμαστε πρόοδο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής Προεδρίας, αλλά επίσης χρειαζόμαστε να εξασφαλίσετε εσείς ως Πρόεδροι ε, ότι τα κράτη-μέλη θα αποφύγουν στο ενδιάμεσο να λάβουν μονομερή μέτρα. Γιατί ήδη η εσωτερική αγορά είναι κατακαιρματισμένη και αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στο πακέτο κινητικότητας και στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά το Brexit. Όλοι γνωρίζουμε το πώς κινείται η διαδικασία και, πώς, πού βρίσκονται οι ευθύνε, αλλά αν δεν εξασφαλίσουμε μία σημαντική μεταβατική περίοδο, θα έχουμε σημαντικό αντικτυπώ στις επιχειρήσεις, στην οικονομία και γενικότητα στη συνδεσιμότητα. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς όμως ε, ε, την άποψή σας αν θα το έχει λάβετε αυτό υπόψη και πώς. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω ε, και ζητώ ξανά συγγνώμη που ε, θα χρειαστεί να φύγω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κράμερ. Κύριε Υπουργέ, και έξω ονόματο ομάδα των Πρασίνων, φυσικά σα εύχομαι κάθε επιτυχία στην πρώτη Προεδρία του Συμβουλίου που αναλαμβάνει η χώρα σα, η Βουλγαρία. Και θα σα στηρίξουμε όσο μπορούμε. Ένα βασικό ερώτημα είναι ο αθέμτος ανταγωνισμός. Μιλήσατε για τα διόδια και για τη σιδηροδρόμους έχουμε ζητήσει να υπάρχει ένα διόδιο και για τους σιδηροδρόμους με χιλιόμετρική απόσταση στα ε, κράτη-μέλη εναπόκειται να αποφύγουν. Ε, στην ε, περίπτωση των ε, σιδηροδρόμων έχουμε 100% διόδια στους δρόμους 1%. Οι οδικές μεταφορές τελικά ενώ ουσιαστικά μολύνουν το περιβάλλον και είναι επιζήμιες επιδοτούνται κατά κάποιο τρόπο, ε, εποφελούνται. Το αντίθετο συμβαίνει με τις ιδρομικές μεταφράσεις. Ό,τι δεν αφορά και την εσωτερική ναυσιπλοή και την ναυσιπλοή γενικά δεν χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιούνται, ε, χρησιμοποιείται βαρύ πετρελαίο, ε, να παράγω εγώ τις πετρελαίου από, από τα πλοία αυτά. Ε, τα οποία μολύνουν 500 φορές ε, το κλίμα από το πιο βρώμικο ε, διζελοκίνητο όχημα στην Ευρώπη. Τι θα κάνετε λοιπόν με την, με, την χρήση αυτού του καυσίμου στην περίπτωση της ναυσιπλοείας για να έχει μια προοπτική ο τομέας και στην περίπτωση του Δούναβη επίσης και τη στρατηγική υπάρχουν πάρα πολλοί λιγότερα ε, πάρα πολύ μεγάλα πλοία από όσα υπήρχαν πριν 30 χρόνια, 3-4 μόνο, αλλά για την περιοχή είναι σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, πτωχεύει η Air Berlin, ποια είναι τα θύματα, οι επιβάτες που είχαν ήδη κλείσει εισιτήρια ε, και οι αεροπορικές εταιρείες δεν τιμωρούνται. Το αντίθετο πάντα συμβαίνει με τους σιδηροδρόμους. Δεν θα πρέπει να έχουν μια ασφαλιστική κάλυψη υποχρεωτική. Οι εταιρείε αυτές υπάρχουν σαν περίπτωση που πτωχεύσουν. Υπάρχει ένα αποθεματικό ε, και να αναγκάζεται η εταιρεία να πληρώσει αυτά και όχι τελικά να την πληρώνει ο επιβάτης, ο πελάτης και κάτι άλλο μεταξύ Βίντεν και Καλαφάτ, νέα γέφυρα στο Δούναμι. Υποτίθεται ότι αυτό είναι καλό ε, για την Ευρώπη. Έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο, εκεί έχουμε συνδρομικές ράγες ε, και ε, ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η αυτή η περιοχή και για τον ποδηλατικό τουρισμό. 44 συγγνώμη, ε, δισεκατομμύρια ε, ο τουρισμός. Αλλά βέβαια έχουμε και την αυσιπλοεία που ε, δίνει πάρα πολλά περισσότερα. Δεν θα πρέπει να δώσουμε και για τον ποδηλατόδρομο κάποια χρήματα. Πώς θα προχωρήσετε. Έχουμε τον 13, έχουμε τον 6 υπαριθμών ποδηλατοδρόμους. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και τον πολιτιστικό, ε, φυσιοδηφικό οικολογικό τουρισμό. Ε, ελπίζω η Ευρώπη να ευελθεί από την εξάμεινη Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Κύριε Υπουργέ, όπως βλέπετε, λέει πρόεδρος, υπάρχουν πάρα πάρα πολλές ερωτήσεις για εσάς. Αλλά για να σας βοηθήσω θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Οι συντονιστές έκαναν αρχικά πολλές ερωτήσεις για αυτό το πρώτο πακέτο κινητικότητας. Ποια θα είναι η θέση της Βουλγαρικής Προεδρίας. Καμποτάζ. Αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Ποιοι είναι οι στόχοι σας. Πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε για να βρούμε διέξοδο σε όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, πολλά ερωτήματα έγιναν για το Δούναβι Πολλά ερωτήματα έγιναν ε, από τον Ρόμπιν και Ρομπερτ Τσίλε, για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση, για τον προπολογισμό, ε, για τις μεταφορές και για το μηχανισμό ε, διασύνδεση. Ο κύριος Τελίτσκα πήγε και λίγο πιο πέρα, τη συλλογιστική λέγοντας ότι συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση των υποδομών που μιλάτε για μια δήλωση τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Επίσης ο ανταγωνισμός ε, στις ε, νέες μεταφορές. Ξέρουμε πόσο αθέμητος ανταγωνισμός υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Και το Brexit αναφέρθηκε. Γιατί θα βρεθείτε στο επίκεντρο της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω αν σήμερα έχετε κάποια ε, στοιχεία απάντησης να μας δώσετε σε σχέση με τις πίστες εργασίας με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους που βρισκόμαστε και τελειώνω με τον ε, κύριο Μιχάλη Κράμερ που μιλάει για τη χρηματοδότηση των οδικών μεταφορών και όχι των σιδηροδρομικών μεταφορών που όμως χρειάζονται αυτή τη χρηματοδότηση και ε, όλα τα όσα ε, είπε και για την ήπια κινητικότητα ε, και τον ποδηλατόδρομο 6 και σίγουρα ο ποδηλατικός του που είναι πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι συνοψίζω λίγο πολύ αυτά που ρώτησαν οι συνάδελφοι. Θα σας δώσω το λόγο για κανένα δεκάλεπτο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Благодаря, госпожо Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, με τις ερωτήσεις του κυρίου Κράμερ. Ο κύριος Κράμερ έθιξε ένα θεμελιώδες ζήτημα για τις μεταφορές. Όχι μόνο στα κράτη-μέλη ξεχωριστά, αλλά στο σύνολο της Ευρώπης. Και αυτό είναι η φορολόγηση, η δίκαιη φορολόγηση των μεταφορών και όλων των τύπων μεταφορών. Η χρηματοδότηση των μεταφορών αυτή τη στιγμή έχει στρεβλώσεις και χρειάζεται να να φέρουμε μια ισορροπία ξανά στο θέμα αυτό. Σε πολλά κράτη-μέλη τα τέλη συνδέονται όχι μόνο με την συντήρηση των υποδομών αλλά και με άλλους παράγοντες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης των οδικών μεταφορών και διαφορετικά για τις άλλες μεταφορές. Για παράδειγμα, η βινιέτα στις οδικές μεταφορές. Η κυκλοφορία των φορτηγών ε, δημιουργεί μεγαλύτερες ζημίες στις ε, υποδομές και, είναι, και μειώνει την ασφάλεια. Συνεπώς, όταν τα βαρέα φορτηγά φορολογούνται λιγότερο από τα άλλα, δημιουργούνται σημαντικότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των υποδομών. Άλλωστε, τέτοια συστήματα φορολόγησης με χαμηλή φορολογία στα βαρέα φορτηγά πλήττει την δυνατότητα ανάπτυξης υποδομών για άλλου τύπου μεταφορές. Ένα αέριες, διαθαλάσσεις κλπ. Γι' αυτό χρειάζεται να ανακτήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους τύπους μεταφορών και κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κάθε τύπος μεταφοράς πρέπει να, να χρηματοδοτείται με τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός με, τις υπόλοιπες, ε, με, τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Θα πρέπει δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των τελών, διοδίων κλπ. Ο, να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες σχετικοί με το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Η ε, επιπτώση που έχει στις υποδομές, στην ασφάλεια των πολιτών κλπ. θα πρέπει να προωθήσουμε και άλλες μεταφορές, όχι μόνο τις οδικές. Αυτή τη στιγμή τα τέλη για ε, που βαρύνουν τα βαρέα φορτηγά στις οδικές μεταφορές είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις επιβαρύνσεις άλλων τύπων μεταφοράς και σας βεβαιώνω ότι θα εργαστούμε στην διόρθωση αυτής της τρέβλωσης. Θα εργαστούμε έτσι ώστε οι επιβαρύνσεις να είναι δίκαιες και ισόρροπες. Σε ό,τι αφορά τις εναλλακ... τους εναλλακτικούς τύπους ε, κινητικότητας, την, ε, ε, το ποδήλατο για παράδειγμα, και τις αντίστοιχες υποδομές με ποδηλατόδρομους. Είναι μια πολιτική προφανώς αυτή που αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Όταν όλοι, όλα τα μέσα μεταφοράς αρχίσουν να επιβαρύνονται με δίκαιο τρόπο, τότε θα αυξηθεί η χρήση των εναλλακτικών τύπων μεταφοράς. Μας δόθηκε το παράδειγμα της γέφυρας πάνω από το Δούναβι ε, μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Εκεί, για παράδειγμα, προβλέπεται και ποδηλατόδρομος. Συνεχίζουμε την ερώτηση για το Brexit. Θα αναφέρω τα λόγια του Πρωθυπουργού μας. Πρόκειται για ένα διαζύγιο και όπως οι όλες οι οικογένειες αυτοί που πιο πολύ υποφέρουν από, το, από ένα διαζύγιο είναι τα παιδιά. Δική μας ευθύνη είναι να βρούμε ένα τρόπο που θα επιτρέψει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσουν φιλικές διμερείς σχέσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, έχουμε ένα ζήτημα με τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Έχουμε τις ε, διαφωνίες μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου για το Γιβλαρτάρ Και αυτά τα δύο ζητήματα μας δυσχεραίνουν. Το Συμβούλιο βέβαια θα έχει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης αλλά αμφιβάλλω για το κατά πόσο για παράδειγμα το Γιβλαρτάρ μπορεί να ρυθμιστεί ε, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά το Γιβλαρτάρ εξακολουθεί να είναι το βασικό πρόσκομα στις διαπραγματεύσεις για τον ε, νέο ευρωπαϊκό ουρανό μετά τον Brexit. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τις οικονομικές και άλλες διμερείς σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά τρία μπλοκ είναι ήδη έτοιμα το ένα από αυτά αφορά εμάς και τη Ρουμανία. Η ενοποίηση του ενέργειου χώρου μας ε, μας επέτρεψε να κάνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα του πακέτου για τις ε, ε, εναέριες μεταφορές και την αεροπλοεία. Πιστεύω ότι θα γενικευθεί ε, αυτή η τάση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σιδηροδρομικές μεταφορές. η χρηματοδότηση των υποδομών γίνεται με χρηματοδοτικά εργαλεία όλο και πιο εξελιγμένα, όλο και περισσότερο ε, προσφεύγουμε σε ελαστικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα την ε, πρωτοβουλία συνδέοντας στην Ευρώπη και άλλου τύπου ε, χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε και τους μηχανισμούς συνοχής. Θα πρέπει όταν δαπανούμε χρήματα των φορολογουμένων μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί Οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ όμω θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Ε, να μην απαιτούμε δηλαδή ε, άμεση κερδοφορία. Θέλουμε η πολιτική συνοχής να παραταθεί σε ό,τι αφορά το πακέτο ε, κινητικότητας και ιδιαίτερα στο πρώτο πακέτο, ακούμε τους πάντες Βέβαια, οι θέσεις των κρατών μελών απήχαν πολύ μεταξύ τους, αρχικά. Σήμερα, όμως, θεωρώ ότι για το πρώτο πακέτο μπορούμε να πετύχουμε σύγκληση. Έχουμε πλέον επικοδομητικές προτάσεις συμβιβασμού από κάποια κράτη-μέλη και αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Σε ό,τι αφορά την οδηγία απόσπαση οδηγών, επαγγελματιών οδηγών, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν θα είναι εύκολο να συγκλίνουν οι απόψεις των κρατών μελών που πολύ συχνά ε, κινούνται προς τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχω ακούσει εκπροσώπους διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων, μεταφορέων στην Ευρώπη και το συμπέρασμα μου είναι ότι οι επιφυλάξεις τους δεν αφορούν τόσο πολύ το... τον πολιτικό χαρακτήρα των προτάσεών μας, αλλά τον τεχνικό, τις τεχνικές πτυχές. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό. Έτσι θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία διαδρόμων και την σύνδεση με τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Εδώ έχουμε δύο διαδρόμου τον υπαριθμόν 8 που ξεκινάει από την Ιταλία, περνάει από την Αλβανία, μετά από τη Μακεδονία, λέει ο μιλητή, και τη Βουλγαρία. Και ο δεύτερο διάδρομο είναι ο 10 που αποτελεί σύνδεση με τη Σερβία. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει. Τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ε, έχουν δικαίωμα να προσδοκούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς όλη η περιοχή θα αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλούμε για προοπτική ένταξης αύριο. Έτσι. Ούτε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Κομισιόν όμως πρέπει να δώσουμε σε αυτές τις χώρες μία ε, μεσοπρόθεσμη ε, προοπτική. Και οι υποδομές μεταφορών είναι μία πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία να εντάξουμε αυτές τις χώρες στο χάρτη της προσβασιμότητας. Σε ό,τι αφορά τον να θα πρέπει να βρούμε μέσω δημοπράτησης μια οδηγία, μια εταιρεία που θα ε, αναλάβει το έργο θα πρέπει να συνδυαστούμε με τους Ρουμάνους διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία είναι αλληλοαποκλειούμενα. Το σύστημα βυθοκόρησης που έχει επιλέξει μία χώρα είναι διαφορετικό από αυτό της άλλης. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία, κατασκευή μάλλον, πρόσθετων γεφυρών Ανάλογα με το ποιο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί και θα έλξει περισσότερους, προσελκύσει μάλλον, περισσότερους επενδυτές, θα δούμε ποιο θα είναι και το μέλλον του Δούναβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε περισσότερη ώρα γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ένα με ένα μισή λεπτό οι υπόλοιποι για να είστε αποτελεσματικοί. Η κυρία Ρεβόνταλόν έχει το λόγο. Ένα με ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μάθω για το πακέτο κινητικότητα σχετικά με την τιμολόγηση. Θέλετε να καταλήξουμε ε, στην ε, ευρωπαϊκού τύπου χρέωση μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Πώς βλέπετε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συγκεκριμένη οδηγία και για την απομάκρυνση από το σύστημα των Eurovignet. Και τι πιστεύετε για την πρόταση την οποία έχω κάνει έτσι ώστε τα έσοδα να στραφούν στις υποδομές μεταφορών. Για το θέμα τώρα το κοινωνικό είπατε ότι ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να υπάρξει σε επίπεδο κρατών μελών. Στόχος αυτού του πακέτου είναι να καταλήξουμε σε ένα κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα υπάρξει ο διάλογος αυτός ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και συμβιβαστική πρόταση για τον κανονισμό σχετικό με την πρόσβαση στην αγορά μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζει την υποχρεωτική ανάπαυση των 45 ωρών στην καμπίνα, πώς θα το απαγορεύσετε αυτό, τι μέτρα θα πάρετε. Και στον τομέα του ανταγωνισμού στις ε, αερομεταφορές, πώς θα προσπαθήσετε να διευκολύνετε ε, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες. Η κυρία Λουκασένσκα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Βουλγαρική Προεδρία έρχεται σε μια δύσκολη φάση. Συζητάμε το πακέτο κινητικότητας, συζητάμε τα θέματα του Brexit. Η συγκυρία είναι δύσκολη, εύχομαι όμως να ισορροπήσετε την κατάσταση και την αποκαταστήσετε την ισορροπία ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση και οι πολίτες να μείνουν ικανοποιημένοι και να κατανοήσουν την ε, προσπάθεια την οποία κάνουμε. Είπατε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις και ότι υπάρχουν και κάποιες εντάσεις σχετικά με το πακέτο κινητικότητας ανάμεσα στις χώρες της Δύσης και στις χώρες της Ανατολής. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι όμως να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά και εδώ οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ δύσκολες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι περισσότερο πολιτικά παρά θέματα ουσίας. Δώσατε αρκετές απαντήσεις για θέματα όπως το καμποτάζ σαν παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει απεριόριστο αριθμό ε, παροχής υπηρεσιών μέσα σε ένα διάστημα πενθήμερο ενώ υπάρχουν άλλες προτάσεις οι οποίες περιορίζουν τη χρονική διάρκεια του καμποτάζου σε δύο ημέρες. Υπάρχει επίσης και το θέμα της μείωσης των εκπομπών που συνδέονται ε, με το καμποτάζ και η ιδέα αυτή μπορεί από ό,τι φαίνεται να ακυρωθεί. Με τους αποσπόμενους οδηγούς θα πρέπει να καλύπτονται από την πρώτη ημέρα και τι γίνεται με την περίοδο ανάπαυσης μέσα στον θάλαμο του φορτηγού τους. Σας ευχαριστώ κυρία Λουκασένσκα. Σταματήσατε κι εσείς περίπου στο 1,5 λεπτό. Η κυρία Φώστερ 1,5 λεπτό πάλι. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τη Βουλγαρική Προεδρία και τον Υπουργό. για την έκθεση για τον ανταγωνισμό. Είμαι μία από τις σκιώδεις της ηγήτρες. Δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για το Συμβούλιο ε, για τα θέματα του ανταγωνισμού, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να ορίσουμε ακριβώς το τι σημαίνει ε, δίκαιος ανταγωνισμός. Το θέμα τίθεται από τη στιγμή που απελευθερώσαμε την, τις αερομεταφορές εδώ και 25 χρόνια και αυτό επέτρεψε να υπάρξει μεγαλύτερη συνδεσιμότητα. Και δεν θα ήθελα να ληφθούν μέτρα τα οποία να θεωρηθούν προστατευτικά και τα οποία να περιορίσουν την ελευθερία της ε, ε, αγοράς των αερομεταφορών στην Ευρώπη γιατί θα αυξήσει ε, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίσης των μεταφορέων από τον υπόλοιπο κόσμο που παρέχουν σωστή συνδεσιμότητα στον κόσμο όλο. Ε, θυμίζω ότι στην Ευρώπη ε, επίσης ε, υπάρχουν κατασκευαστές και ταυτόχρονα γι' αυτό λοιπόν επειδή τα προϊόντα αυτά εξάγονται σε εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Τώρα για το Γιβλαρτάρ δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά το 2006 υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στο Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, στον αερολιμένα του Γιβλαρτάρ ε, μη ε, στρεβλές ανταγωνιστικά πρακτικές. Δεν ε, είναι το θέμα τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε ε, το τι είναι κυρίαρχο έδαφος και τι δεν είναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τη Βουλγαρική Προεδρία και εγώ και να σας ενθαρρύνω, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μικρότερες χώρες έχουν καταφέρει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ε, στα χρόνια εδώ που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω την ίδια τύχη να έχετε και εσείς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε ήδη ακούσει πολλά ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά όμω ε, το πρώτο πακέτο, επειδή είμαι εισηγήτρια για την οδηγία με, για την ε, απόσπαση των εργαζομένων και έγιναν κάποιε από τι ερωτήσει που ήθελα και εγώ να σα ε, θέσω, θέλω να σα κάνω μια άλλη ερώτηση Απέναντι στον κίνδυνο, όπω είπατε και εσεί ε, και τι δυσκολίε που μπορεί να προκύψουν για την οδηγία λόγω των κρατών μελών, βλέπετε το ενδεχόμενο ε, να μην ε, περάσει το πακέτο, να σπάσει σε κομμάτια, δηλαδή να προχωρήσουν άλλες μεταρρυθμίσει, άλλε να μείνουν πίσω, γιατί είπε ο Επίτροπος Μπούλτ ότι μόνο αν όλε οι μεταρρυθμίσεις προχωρήσουν ταυτόχρονα έχει σημασία αυτό το πακέτο. Επίση, ότι αφορά τι συνδυασμένε μεταφορέ που αναφέρατε ω έναν από του στόχου, σα είπατε μια οδηγία εμείς έχουμε εγκρίνει την νομοθεσία ε, και το έχουμε κάνει και με άλλες οδηγίες. Βλέπουμε όμως ότι δεν τηρείται αυτή η νομοθεσία από τα κρατημέλα, άρα από οργανωτικής πλευράς καταστροφή για την Ευρώπη. Ποιοι θα είναι οι στόχοι στους οποίους θα εστιάσετε σε ό,τι αφορά την οδηγία που προτείνεται για τις συνδεσμένες μεταφορές επί της δικής σας προεδρίας και τέλος υπάρχει μια πρόταση κανονισμού για κοινούς κανόνες ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διεθνή αγορά των πούλμαν και των λεωφορείων. Έχετε ήδη λάβει αρνητικές ε, αναφορές από κάποιες χώρες όπως από την Μικτή Επιτροπή Γερουσίας και Βουλής ε, της Ισπανίας. Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πρόεδρο σας, ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Αλλά παρακαλώ να προσπαθείτε να τηρείτε το χρόνο σας γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις απαντήσεις η κυρία Ταρπαντέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ Μεταφορών και Υποδομών της Βουλγαρίας. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και πραγματικά αποδίδω ύψης της σημασία στο γεγονός πως η Βουλγαρία έχει το εξάμεινο αυτό την εκπεριτροπής προτριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρώτη φορά που μια χώρα που προσφάτως προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται των εργασιών των κρατών μελών. Τρεις πτυχέ. Πρώτον, οι οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες συνδεσιμότητας με την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην έκθεση για την αξιολόγηση της συνδεσιμότητας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχα επιμείνει στο γεγονός αυτό. Η περιοχή αυτή έχει ιδιαιτερότητες, άρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη στρατηγική. Άρα αυτό ζητεί περισσότερη τεχνική αλλά και χρηματοοικονομική ενίσχυση από πλευρά κομισιών. Θα πρέπει επίσης ε, να επιβεβαιωθούν τα σχέδια τουρισμού και επενδύσεων. Συμφωνεί η Βουλγαρία. Προβλέπει δράσεις για να στηριχθούν αυτές οι στρατηγικές ανάπτυξη κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης τώρα. Ναυσιπλοεία, αστέρια σου στο Δούναβι είναι ένα λεπτό ζήτημα, πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρουμάνια και τη Βουλγαρία. Πάνω από 500 χιλιόμετρα του ποταμού αυτού ε, τα μοιραζόμαστε δύο χώρες, Βουλγαρία και Ρουμανία και αυτό είναι σημαντικό για τις χώρες μας αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πράγματι, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τη βεθοκόρηση υπάρχουν α, ίσως διαφωνίες. Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δύο υποδομές. Υπάρχει όμως καθυστέρηση και χρονοτριβή και αυτό επηρεάζει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μέσω του Δούνευ. Για το χώρο Σέγγεν τώρα θα ήθελα την επιβεβαίωση ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα έχουν μια κοινή στρατηγική για να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν. Γιατί όμω το θέτω εδώ το ερώτημα στην Επιτροπή Μεταφορών, γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Όμω αυτό πλήττει τι εμπορευματικέ ε, μεταφορέ και την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Τζαμπάσκι. Τζαμπάσκι, καλά σας πρόφερα το όνομα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ. Δεν θα έχετε εύκολο εγχείρημα ως υπουργό επί Βουλγαρικής Προεδρίας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών, όπως είδατε, είναι άκρος δραστήριοι και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το ζήτημα της απόσπασης των οδηγών. Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ συνήθω έχουν να κάνουν με την γεωγραφία, διότι κάποια κράτη-μέλη έχουν κάποιες εντάσεις, Σλοβανία, Σλοβεκία, Εστονία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Το καμποτάζ επίσης είναι ένα δύσκολο θέμα. Είναι ένας τομέας όπου δεν υπάρχει ευρωπαϊκός οργανισμός. Υπάρχει ένας οργανισμός για τις ενέργειες ε, μεταφορές, για τις θαλάσσιες μεταφορές, όχι όμως για τις οδικές. Διερωτώ με λοιπόν κατά την άποψή σας. Και έχοντας υπόψη το Brexit και τη βούληση μείωση των δαπανών. Θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο οργανισμό, τι πιστεύετε. Θα ήθελα επίσης τι, θέλετε, τι μπορείτε να μας δείτε και τα τηλεδιόδια στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ε, καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ. Άκουσα με πολύ προσοχή την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για τη διεύρυνση, και υπό την προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Εξήγησε ότι η Βουλγαρία θα στραφεί και προς ε, τα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ είμαι και Σέρβος υπήκος και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσέγγιση με αυτή την περιοχή. όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορούν ε, οι πολιτισμοί να έρθουν πιο κοντά, αν δεν έρθουν πιο κοντά και τα κράτη. Η Βουλγαρική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες ε, της κοινότητας μεταφόρων των Βαλκανίων. Ξέρετε ότι έχει συναυθεί και μια συμφωνία μεταξύ των χωρών αυτών υπό λοιπόν, την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την κοινότητα. Η οποία πλέον είναι πραγματικότητα. Θα επωφεληθείτε από αυτή τη νέα οργάνωση. ώστε να δοθεί όθηση στις μεταφορές και στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Είμαι εισηγητής ε, του Lex Specialis για την απόσπαση από το ΕΛΚ και επειδή εξηγήσατε ότι κατά τη δική σας άποψη είναι ένα λεπτό θέμα, θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξο. και αν θα προσπαθήσετε κι εσείς να βοηθήσετε να δοθεί μια γενική κατεύθυνση, ένας γενικός προσανατολισμός στο εξάμεινο της Πρόεδρες σας. Ευχαριστούμε κυρία Ντελμόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι καλύτερες ευχές μας προς την Βουλγαρική Προεδρία. Θα μιλήσω ειδικά για τα Βαλκάνια με αφορμή την Ολομέλεια και μια παρέμβαση την οποία είχα κάνει πρόσφατα για το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει σημασία και πρέπει να τίθεται συνεχώς. Σαν Επιτροπή Μεταφορών λοιπόν Ενδιαφέρομαι για να λειτουργήσουν τα TNT, να υπάρξουν επενδύσεις και σε σχέση με τον δρόμο του μεταξιού και για τη βελτίωση των υποδομών μεταξύ των οποίων και των λιμένων. Πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δικτύων TNT και στα Βαλκάνια. Αναφερθήκατε στη συνάντηση κορυφής στη Σόφια και γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και μια συνάντηση κορυφής η οποία θα εντάσσεται στα πλαίσια της διαδικασίας του Βερολίνου. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν εμπλέκεται στα στάδια αυτά. Εσείς θα υποστηρίξετε τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής. Σόφια και Βερολίνο και εδώ έρχομαι να συμφωνήσω με τον συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα, πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την κοινότητα των μεταφορών, κύριε Ντεμόντε. Ο κύριος Κούνι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Σας καλωσορίζουμε στις μεταφορές και ο τομέας των μεταφορών και των υποδομών είναι ε, πράγματι πολύπλοκος. Έχουμε και το θέμα του τουρισμού. Η Βουλγαρία είναι μια υποδεχματική τουριστική ε, χώρα, η αρένα, ε, η παραλία αυτή και άλλες ακτές και έχουμε και το θέμα ε, της ε, οικονομίας και οικολογίας όταν αυτά δεν συμβαδίζουν. Άκουσα από τον Πρωθυπουργό γιατί ρωτώ τι θα γίνει αλλά, ε, με το τελεφερικ, αλλά δεν ξέρω πώς ε, αντιλαμβάνεστε τον οικολογικό απολογισμό των διαφόρων έργων για τις μειώσεις των εκπομπών καυσαερίων πρέπει να βλέπουμε γενικά τα πράγματα ε, για τους αυτοκινητοδρόμους, ε, για τα διόδια, τηλεματική. Ε, δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις. Πώς θα τις επιλύσετε εσείς ε, ως Υπουργός Μεταφο... Υποδομών. Συγγνώμη με την κυρία Γιάλα Σέντερ, ενάληψη λεπτό. Μην το υπερβείτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, απλά θέλω να σας πω ότι σύντομα επί Προεδρία σας θα κατατεθεί από την πρώτη πρόταση ε, για τον προπολογισμό ε, στο, του μέλλοντος Ευρώπης, ε, τρίπλο κονδύλια για τον ορίζοντα 2020, για την άμυνα, πολλά περισσότερα κονδύλια κτλ. Μας ανησυχεί λοιπόν όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ τι θα γίνει με τον προπολογισμό για τις μεταφορές στο πλαίσιο του Connecting Europe μήπως δεν υπάρξει βελτίωση ε, στον επόμενο προπολογισμό. Έχετε σκεφτεί ε, στην Προεδρία σας εσείς ε, κάποιο πρόγραμμα, κάποια δήλωση και για το πακέτο και για την κινητικότητα. Η Προεδρία σας ίσως καλό θα ήταν να τόνιζε ή να έδινε έμφαση σε ένα πακέτο κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Γιατί ένα πρόβλημα που έχουμε και εκεί πρέπει να δοθεί απάντηση είναι ότι έχουμε τα φορτηγά με τόσες πολλές υποχρεώσεις ευθύνε και παίρνει και όλο το φταίξιμο σε οδικές μεταφορές, αλλά τι γίνεται με τους ελέγχους. Συχνά βλέπουμε διακριτική μεταχείριση. Δεν πρέπει οι φορτηγατζίτες να μπλοκάρονται, και για τις τιμές ε, των μεταφορών και των ε, αρχών φόρτωση εκφόρτωση. Γιατί υπάρχουν οι τιμές των προϊόντων που επηρεάζουν και όχι απλά ε, τα φορτηγά. Λοιπόν, τώρα στρέφαμε στον κύριο Υπουργό. θα πρέπει να προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για αυτό που ονομάζουμε Ευρωβινιέτε, τι το ευρωπαϊκό τέλος. Ε, η, η, συγκεκριμένη στόχευση των εσόδων από, από τα έσοδα, ή μάλλον ένα τμήμα τουλάχιστον για συγκεκριμένους στόχους κοινωνικούς ή θέματα υποδομών. Ο κοινωνικός διάλογος επίσης, πώς ακριβώς θα προχωρήσετε. Η... Αν μπορούσατε να αφήσετε τον Υπουργό να απαντήσει μόνος του χωρίς να επαναλαμβάνετε και να ερμηνεύετε τις ερωτήσεις μας, αν επιτρέπετε. Ας απαντήσει ο Υπουργός. Κυρία Σέντερ, ο στόχος είναι να τον βοηθήσουμε. Κάνω μια σύνοψη των ερωτήσεων για να ε, βοηθήσουμε τον Υπουργό. Ε, ο κάθες από εσά έθεσε περισσότερα από ένα ερωτήματα, δύο, τρία, οπότε προσπαθώ να βοηθήσω τον Υπουργό, δεν προσπαθώ να αλλοιώσω τι ερωτήσει σα. Όταν γίνεται ε, λόγος για το, τα θέματα των διαλυμάτων και των ανάπαυση των οδηγών. Αυτό, για παράδειγμα, ετέθη από, και από την κυρία Μπιλμπάου. Ε, οπότε, εγώ τα συνοψίζω. Συνδυασμένε μεταφορέ μετά. Πραγματική ερώτηση. Καλή ερώτηση. Ποια θα είναι η θέση σας για, την, ε, για τα πούλμαν και τα λεωφορεία και τις μεταρρυθμίσεις αυτά. Μετά, η θέση των Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό ε, πανόραμα μεταφορών. Ο κ. Τζαμπάσκι έθεσε το ερώτημα που θέσατε και εσείς κυρία Γιάλα Σέντερ. Είστε υπέρ ή κατά μιας υπηρεσίας. Λέει, κάτι λέει για το Σέντερ, κυρία γιαννα Σέντερ, εκτός μικροφώνου. Και Τέλος, ε, τα θέματα του προπολογισμού των ε, μεταφορών, πώς μπορεί να ε, αυξηθεί ο προπολογισμό με ποιο τρόπο κλπ. Τώρα, δίνω το λόγο σε εσά κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Και οι δικοί μου βοηθοί προσπάθησαν να μου τα ομαδοποιήσουν. Στηρίζουμε την δημιουργία μιας ειδική υπηρεσίας ελέγχου και καθορισμού κανόνων για τις οδικές μεταφορές. Ε, ένα σύστημα ενιαίας τιμολόγησης των οδικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει ένα καλό βήμα προς το μέλλον. Ένα τέτοιο σύστημα θα κάνει πολύ καλό στην τομέα των μεταφορών, αλλά θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνον αν οι οδικές μεταφορές ε, ε, ε μέσα σε ένα πλαίσιο με τους άλλους τύπους μεταφορών. Περνάω στις άλλες ερωτήσεις. Ευρωβινιέτα. Στηρίζουμε την, το στόχο αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή να γίνει σεβαστή αρχή να γίνουν σεβαστές οι αρχές ορυπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Το σύστημα της Ευρωβινιέτας θα πρέπει να ωφελεί τον Ευρωπαίο πολίτη και σκοπεύουμε να κάνουμε ένα απολογισμό το, της πρόοδου που έχει επιτευχθεί με στόχο να διαθέτουμε στα χέρια μας μια στέρεη βάση για την διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών. γνωρίζουμε τις διαφορετικές απόψεις. Θα προωθήσουμε ένα λειτουργικό, βιώσιμο ε, και δίκαιο τομέα κλάδο μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα τόσο των επαγγελματιών οδηγών όσο και τα οικονομικά συμφέροντα των μεταφορέων. Οι αποφάσεις ε, όμως, οποιασδήποτε αποφάσεις δεν θα πρέπει να αυξήσουν την γραφειοκρατία. Θα πρέπει να βασίζονται επίσης σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Σε ό,τι αφορά το καμποτάζ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διεθνών οδικών μεταφορών. Στόχος είναι να περιορίσουμε τον αριθμό των, ε, της, ε, των φορτηγών που κινούνται άδεια και ένα φορτίου, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Θέλουμε να... Ε, ο οποιοδήποτε καποτάζ γίνεται να γίνεται σε, με τη, επί τη βάση νομιμότητας με αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί, πιστεύουμε, βελτιώνοντας τις τεχνολογικές πτυχές του. Με ευφυείς ταχογράφους, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Η κοινωνική πτυχή συνδέεται με την εμπορική πτυχή του πακέτου και γι' αυτό το λόγο αυτές οι δύο θα πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευσης ε, παράλληλα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τις πτυχές που είναι πιο συνενετικές και μετά να περάσουμε στις άλλες η επεξεργασία κανόνων ε, κατά των επιχειρήσεων βιτρίνα ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνει και ε, οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις χώρες οποίες γίνεται το αδίκημα. Η σύνδεση ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο πακέτο κινητικότητας. Η αναδιατύπωση της οδηγίας ε, των συνδυασμένων μεταφορών συνδέεται άμεσα με ζητήματα του πρώτου πακέτου κινητικότητας. Για παράδειγμα, συνθήκες εργασίας και αποσπάσεις οδηγών. Θέλουμε σαφείς κανόνες για τις συνδυασμένες μεταφορές και ιδιαίτερα για το καμποτάζ. Όλοι γνωρίζουμε την εκμετάλλευση την οποία υφίστανται πολλές φορές εργαζόμενοι στο μέτρο των μεταφορών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε την ε, εξέλιξη του τομέα με τρόπο ανταγωνιστικό και βιώσιμο. Θα πρέπει όμως να βρούμε και μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων αφενός και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών αφετέρου. Στηρίζουμε επίσης την δημιουργία μιας ειδική υπηρεσίας που θα χειριστεί τα θέματα ε, κανόνων και ελέγχων για τις οδικές μεταφορές. Και απαντώντας την κυρία Ντέλη, ε, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Είμαι μάλλον σκεπτικός ε, και επιφυλακτικός. Το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό με του συναδέλφους και έχω αντιληφθεί ότι έχουμε βαθιές διαφορές μεταξύ μας. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο για αυτό το θέμα. Αν ξέχασα κάτι, μου το λέτε. Η δική μου ομάδα είναι πιο αισιόδοξη από ότι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ταχύτατος καταφέρατε σε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ξέρω δεν ήταν εύκολο. Αν, δεν έχετε, αν έχετε άλλες ερωτήσεις, γραπτός παρακαλώ στην ομάδα του Υπουργού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιέρωσατε αυτό το χρόνο. Σας, σας περιμένουμε να επιστρέψετε. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συνεργασία μας. Thank you very much. Mes chers collègues, avant de partir, on me signale que pour... Για να έχουμε χρόνο συζήτησης, παρόλο που πολλοί ξεπερνούν το χρόνο τους, θα ξεκινήσουμε το απόγευμα στις 2.30. Στις 2.30. Έτσι. Ευχαριστώ.